Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε τις εργασίες μας. Si veut bien regagner... Euh, καθίστε, σας παρακαλώ, ή όσοι δεν είναι να καθίσετε, βγείτε, παρακαλώ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους για την επανάληψη των εργασιών μας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ελπίζω όλοι να υποφεληθήκατε για να γεμίσετε ενέργεια, να ξεκουραστείτε και να αρχίσετε τη νέα θητεία με την απαιτούμενη δύναμη. Πριν δώσω το λόγο στην Υπουργό κυρία Λάρσον και σας ευχαριστώ που ήρθατε, ήθελα απλά να πω στους συναδέλφους ότι θα γίνει μία μόνο αλλαγή στην ημερήσια διάταξη Πρόκειται για την οργάνωση του χρόνου εργασίας ε, των εκτελούντων εκκίνητές δραστηριότητες ε, οδικών μεταφορών. Είχε προβλεφθεί αρχικά να συζητήσουμε το θέμα και να ψηφίσουμε αύριο. Αλλά θα γίνει μια συζήτηση το απόγευμα και θα αναβάλουμε την ψηφοφορία. Δεν θα γίνει αύριο. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως στο σημείο 4 της μερίσιας διάταξης και θα επανέλθουμε στη συνέχεια σε ό,τι εκκρεμεί. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που ήρθατε. Είστε η πρώτη μας ε, προσκεκλημένη στη νέα θητεία. Ε, είστε αρμόδια για τα θέματα δημόσιας υγείας ε, και για την τρίτη ηλικία. ήθιστε στο Κοινοβούλιο, όπως ξέρετε, να γίνονται ακροάσεις των Υπουργών ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Με αυτή την ιδιότητα έχετε έρθει σήμερα. Και άλλοι δύο συνάδελφοί σας θα έρθουν αύριο. Με αυτή την ιδιότητα λοιπόν ήρθατε σήμερα, όπως ήθιστε στο Κοινοβούλιο, να σας δώσω το λόγο για 10 λεπτά και δεν ξέρω πόσο χρόνο θέλετε, 10-20 λεπτάκια εν πάση περιπτώσει. Και μετά θα κάνουμε μια ανταλλαγή. Ε, κύριε Χένρι, έχετε διαδικαστικό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου την Υπουργό. Θα ήθελα απλώς ε, να ζητήσω επειδή δεν έχουμε εγκρίνει ακόμα την ημερήσια διάταξη, αν μπορούμε να κάνουμε μια ανταλλαγή μεταξύ των σημείων 6 και 7 της ημερήσιας διάταξης, διότι ο εισηγητής ε, έχει μια υποχρέωση σε μια άλλη επιτροπή μπορούμε να κάνουμε μια ανταλλαγή ε, των σημείων 6 και 7. Ναι, ναι, καταλαβαίνω απλά, ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι στο σημείο 7 έχουμε εξωτερικούς, ε, ε, έχουμε προσκεκλημένους δηλαδή που δεν έχουν σχέση με τις εργασίες της Επιτροπής μας για το σημείο 8 και είναι λίγο αργά τώρα να υποβάλλετε τέτοιο αίτημα, δεν σας δημιουργεί πρόβλημα. Προτείνω να παραμείνει ως έχει η σε διάταξη. Δίνω το λόγο στην κυρία Λάρσον. Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, αλλά άκουσα ότι σήμερα, αύριο το πρωί, συγγνώμη, δεν θα ψηφίσουμε το σημείο που είχε προβλεφθεί στην ημέρησια διαταξή και θα ήθελα να ξέρω για ποιο λόγο δεν θα ψηφιστούν αυτά. Σας ε, προτείνω το θέμα αυτό να <clears throat> το συζητήσουμε να φτάσουμε στο σημείο 7 <clears throat> να μην καθυστερήσουμε τα πράγματα τώρα γιατί ε, θέλω αμέσως να δώσω το λόγο στην Υπουργό. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που ήρθα σήμερα εδώ για να συναντήσω τους βουλευτές της Επιτροπής που έχει τόσο ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων και θα ήθελα να σας συγχαρώ, να συγχαρώ τα νέα, τους νέους βουλευτές. Είναι συναρπαστικές οι εργασίες που σας περιμένουν. Έχω έρθει για να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας στο δικό μου το χαρτοφυλάκιο υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με την περίθαλψη των ηλικιωμένων, θέματα δημόσιας υγείας. Θα έρθουν και οι συνάδελφοί μου, η Κριστίνα Χιούσμα Πέσον, που είναι υπουργό αρμόδια για τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης και ε, ο Σβένο Τολιτορίν, πω από δύσκολα ονόματα που σας λέω και που είναι αρμόδιος για την αγορά εργασίας. Αύριο θα έρθουν αυτοί οι συνάδελφοί μου και μπορείτε να τους κάνετε ερωτήσεις και να συζητήσετε και για ε, αυτά τα ζητήματα. θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, διαδραματίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία σήμερα να σας συναντήσω, να συζητήσουμε για αυτό που μας περιμένουν το φθινόπωρο και να σας καλέσουμε να συνεργαστείτε μαζί μας ε, και ευελπιστώντας ε, να μας υποστηρίξετε για τα ζητήματα που είναι της δικής μου αρμοδιότητας κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας. Μία από τις μεγάλες μακροπρόθεσμες προκλήσεις για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι νέες δημογραφικές τάσεις. Θα έχουμε όλο ένα και περισσότερους ηλικιωμένους σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ζούμε περισσότερο. Αυτό είναι φανταστικό. Δείχνει την επιτυχία του κράτους πρόνοιας. Ε, συνιστά μεγάλη πρόοδο για την κοινωνία μας. Αλλά Μεταξύ άλλων θα διαπιστώσουμε ότι όλο και μικρότερο ποσοστό ανθρώπων έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οπότε θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ολόκληρο το δυναμικό στον τομέα της τη Ευρωπαϊκής Ένωσης με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, τόσο ώστε να διατηρήσουμε αυτή την ευημερία που επικρατεί στην Ένωση ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε το μέλλον των ηλικιωμένων και να κατοχυρώσουμε μία αξιοπρεπή και ποιοτική περίθαλψη αυτό συνιστά ένα από τα βασικότερα καθήκοντα που καλείται να υπομειστεί η κοινωνία μας. Η περίθαλψη ε, και το κράτος πρόνοιας για τους ηλικιωμένους ε, θα συνεπάγονται λένε και μεγαλύτερες δαπάνες και επίσης ε, χρειάζεται και να αναβαθμιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών. Αυτό είναι το υπόβαθρο και έτσι επέλεξα να αναδείξω σε προτεραιότητες διάφορα ζητήματα το πιο σημαντικό είναι η αξιοπρεπής και υγιής γύρανση του πληθυσμού. Και θα ήθελα αυτό το θέμα να εγγράφεται στη μερίσια διάταξη Ευρωπαϊκής Ένωσης με πιο μόνιμο τρόπο. Θέλουμε να υπάρχει καλή ανταλλαγή ε, εμπειριών και βελτίστων πρακτικών ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε αυτό το τομέα. Ένα βασικό ζήτημα που θα μας απασχολήσει σε αυτό το τομέα είναι η ανάγκη που υπάρχει να ενισχυθεί η συνεργασία και ο συντονισμός ανάμεσα στον τομέα της υγείας και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης σχετικά με την περίπτωση περίθαλψη και την πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Ε, αυτό θα συνεπάγεται ε, μεγάλα κέρδη, θα αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής ε, για τους ηλικιωμένους και επίσης θα εξοικονομήσουμε και χρήματα. Ε, αυτό είναι το συμφέρον της κοινωνίας. για να έχουμε μια αξιοπρεπή περίθαλψη και πρόνοια για τους ηλικιωμένους πρέπει να αλλάξουμε την, το σημείο εστίασης, δηλαδή να βασιζόμαστε, να έχουμε ως γνώμονα τις ατομικές ανάγκες. Ε, και αυτό η, η περίθαλψη είναι πάρα πολύ σημαντική για όσους δεν μπορούν να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Πάμε μας φέρει κάποιος που πάσχει από Αλσχάιμερ ή από μια άλλη νευροεκφυλιστική νόσο. Ε, αυτές οι ασθένειες πλήττουν όχι μόνο τους ηλικιωμένους αλλά και τις οικογένειές τους και τους συγγενείς τους. Ε, τέτοιες ενώσεις δημιουργούν πολύ συγκεκριμένε απαιτήσει για τη συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και καλούν οι αρμόδιοι να απομεστούν τις ευθύνες τους. Ε, γυράσκει λοιπόν ο πληθυσμό, και αυτό είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολλές προηγούμενες προεδρίες και έχει προεξάρχουσα θέση στο κοινό πρόγραμμα που εγκρίναμε από κοινού με την Γαλλική και την Τσεχική Προεδρία. Θα αρχίσουμε τις εργασίες του φθινοπόρου με μια διάσκεψη ε, στη Στοχόλμη στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου ε, θα έχουμε προσκαλέσει εμπειρογνώμονε και πολιτικού παράγοντε από τα κράτη-μέλη, από τα θεσμικά όργανα τη Ένωση και από διάφορε οργανώσει για να γίνει ανταλλαγή εμπειριών και βελτίωση των πρακτικών για να δούμε πώ μπορούμε να προάγουμε ε, στο μέλλον ε, την κοινή δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι πάρα πολύ που θα υπάρξουν και βουλευτέ. σε αυτή τη διάσκεψη που διορθώνει οι διερμηνέ είναι στι 15 και 16 Σεπτεμβρίου. Ε, η φιλοδοξία μας είναι στην 1η Δεκεμβρίου θα γίνει το Συμβούλιο ΕΦΚΟ, αν δεν κάνω λάθος, θα εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με την αξιοπρεπή και την ενεργό γύρενση. Ο στόχος μου είναι αυτά τα συμπεράσματα συμπεριλαμβάνουν ένα μήνυμα από το Συμβούλιο σχετικά με το πώς μπορούμε να προάγουμε την αξιοπρέπει αξιοπρέπεια συγγνώμη, των ηλικιωμένων και την ποιότητα ζωής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο δράσης για να αναλυφθούν μέτρα σε επίπεδο ένωσης, ούτως ώστε να υποστηρίξουμε αυτού τους στόχους. Ένα σημαντικό μέτρο θα μπορούσε να είναι να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα, ένα κόμβο για να ανταλλάσσουμε εμπειρίε και καλά παραδείγματα ανάμεσα στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου καλούμαστε να ταπεξέλθουμε και στην οικονομική κρίση που μας πλήττει και θα πρέπει να δούμε πώς, ε, τι επιπτώσεις έχει η οικονομική κρίση στον κοινωνικό τομέα. Επίσης, ε, στις εργασίες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα σημειωθούν πολύ σημαντικές αλλαγές ε, στην επόμενη, στο επόμενο εξάμεινο η Ισπανία που θα αναλάβει την Προεδρία έχει ως στόχο να υιοθετηθεί μια νέα στρατηγική για την ανάπτυξη και για την απασχόληση. Ένα σημαντικό σημείο αναφοράς θα είναι η στρατηγική της Λισαβόνας για ό,τι κάνουμε γενικώ στον κοινωνικό τομέα. Ακόμη και πριν από την κρίση Ε, είχαμε ένα ευρύ πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το αποκλεισμό, Σχεδόν 100 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας. Ε, με την κρίση τώρα ε, ενδέχεται να αυξηθεί αυτό το ποσοστό και οι αποκλεισμένοι ε, ενδέχεται να αποκλειστούν ακόμη περισσότερο, να απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από την αγορά εργασία. Για να παρεμποδίσουμε αυτή την εξέλιξη θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. Όταν λέω εμείς τα κράτη-μέλη και υπό υπογαλλική Προεδρία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνουμε μια στρατηγική για να αυξήσουμε την συμμετοχή των ανθρώπων που είναι και οι πλέον ευπαθεί, αν θέλετε στην κοινωνία μα. Ε, ονομάστηκε Active Inclusion Strategy, δηλαδή στρατηγική ενεργού εμπλοκή αυτών των ανθρώπων. Ε, ε, θα γίνει επίσης ένας γύρος τραπέζι 15 και 16 Οκτωβρίου το, το, το, τώρα το φθινόπωρο για την ε, φτώχεια και για τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ε, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός στην καταπολέμηση της φτώχειας, στα πλαίσια της στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις για την ενεργό συμμετοχή θα εστιάσουμε τις συζητήσεις στον τρόπο με τον οποίο αυτή η στρατηγική μπορεί να υποστηρίξει, να επικουρήσει τα κράτη-μέλη ε, κατά την επίρρωση της ε, κοινωνικής συμμετοχής και την καταπολέμηση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Η καταπολέμηση της φτώχειας είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συνεχίσει να συνιστά προτεραιότητα στην μερίσια διάταξη Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το ίδιο, όπως και οι στόχοι για την ανάπτυξη και για την απασχόληση. Από κοινού αποφασίσαμε ότι του χρόνου, ε, θα, μάλλον ε, το 2010 θα είναι η χρονιά της καταπολέμησης της ευτόχειας. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Και σε αυτή την διάσκεψη τρογγυλής τράπεζας υπάρχει ένας άλλος σημαντικός στόχος στόχος, ε, αυτός ακριβώς του 2010, που θα είναι το έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας ε, και ε, νομίζουμε ότι θα γεμίσουμε έτσι με ενέργεια για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας για μεγάλο χρονικό διάστημα στον τομέα αυτό. Ε, τώρα, θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις ε, χρησιμοποιώντας την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, μιλώντας για την κοινωνική ασφάλεια και την κοινωνική συμμετοχή και για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας. Επίσης, αυτή τη διάσκεψη θα λύσουμε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την συνέχεια των εργασιών μας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας από τους σημαντικούς εμπλεκόμενους φορείς που έχουν προσκληθεί ε, να συμμετάσχουν στην στρογγυλή αυτή τράπεζα για να καταλήξουμε τελικά σε κοινά συμπεράσματα. Η πολιτική μας για τα άτομα με αναπηρίες τώρα είναι ένα από τα ζητήματα που αναδεικνύονται σε προτεραιότητες για τη Σουηδική Προεδρία. Το θέμα της πρόσβασης δεν μπορεί να ε, θεωρηθεί ως ένα ξεχωριστό ζήτημα γιατί είναι μία από τις προϋποθέσεις για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα υγιούς και εξευρεπού γύρανσης ε, γιατί οι διάφορες αναπηρίες ε, αυξάνονται όσο ε, μεγαλώνει κανείς. Και η στρατηγική για την ε, ενεργό συμμετοχή είναι πολύ σημαντική για τα άτομα με αναπηρίες και η πρόσβαση είναι ένα θέμα που απασχολεί ως προς όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες που θα επιτελέσουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Δηλαδή σε όλες τις συνεδριάσεις η συνολική η γενική ετικέτα είναι πρόσβαση, ανοιχτή πρόσβαση. Ε, και όπως σας είπα, ε, η η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το τομέα δεν είναι η υποχρεωτική νομοθεσία. Ε, ε, βασιζόμαστε στη βούληση και στη δέσμευση που αναλαμβάνουν και τα κρατη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και οι εμπλεκόμενοι λοιποί φορείς. ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η μερίσια διάταξη για το φθινόπωρο εστιάζοντας στις κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, στην κατάσταση των ηλικιωμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ε, μορφές, ε, της μεθόδους για να συνεχίσουμε την συνεργασία για τα κοινωνικά ζητήματα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά μπορούν να ε, δημιουργήσουν την βούληση και τη δέσμευση που χρειαζόμαστε ούτως ώστε να τελεσφορήσουν οι προσπάθειές μας. Ελπίζω να κάνουμε μια επικοδομητική και ενδιαφέρουσα συζήτηση για αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup. Euh. Και εμείς σας ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε για αυτή την παρουσίαση ενός προγράμματος Σουηδικής Προεδρίας και φιλόδοξου αλλά και ρεαλιστικού αν θέλετε. Φαίνεται ότι ξέρετε καλά την κατάσταση. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συζήτηση, περιμένουμε να ακούσουμε ερωτήσεις. Ο η κυρία Ελίζα Βετλίν, την πρώτη μας αντιπρόεδρος, θα πάρει το λόγο πρώτη και μετά η κυρία Χίλιτα Φιγκερέιρο. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλήσατε για την ενεργή συμμετοχή και ένταξη και για την αναπηρία και για την, τους ηλικιωμένους. Αυτά είναι όλα θέματα για τα οποία ε, συνεχώς φωνάζουμε τα τελευταία χρόνια για το άρθρο 13 του σχετικού πακέτου κτλ. Εγώ θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω τι θα κάνετε συγκεκριμένα για να προωθήσετε ακριβώς το άρθρο 13 της μη διακριτικής μεταχείρισης σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα που ανέφερα. Δεύτερο ερώτημα, οι βέλτιστες πρακτικές και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφορών κρατών μελών για την ε, ε μεταχείριση των ε, κακομεταχείριση των ηλικιωμένων ε, σχετικά μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα και το τρίτο ερώτημα μου σχετίζεται με τα αντιβιωτικά οι στόχοι ας πούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την καταπολέμηση ή τη μείωση αν θέλετε των κρούσματων MRSA που είναι ενδοκοσυ... ενδονοσοκομιακές λοιμόψεις ε, ξέρω ότι στο Ηνωμένο, στο, στη Σουηδία δεν υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό κρούσματων. Μπορείτε να μας πείτε τι θα κάνετε. Πρόεδρος, η κυρία Χίλτα Φιγκερέιδο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, Υπουργέ, για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα ήθελα να θέσω τρεις ερωτήσεις, πολύ σύντομες. Πρώτον, με την επιδείνωση της ε, κοινωνικής κατάστασης λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, έχει ε, επιπτώσεις ε, κυρίως σε δύο ε, μάλλον σε δύο ομάδες, τις γυναίκες και κυρίως τι ηλικιωμένε γυναίκες και ε, ε, στο σύνολο των ηλικιωμένων και των ανέργων. Οπότε τίθεται το εξή ζήτημα. Εφόσον μιλάμε για ενεργό ένταξη και καταπολέμηση της στόχιας, ε, ε, ερωτώ πώς θα ε, αντιμετωπίσετε συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένα για τον κοινοτικό προϋπολογισμό για του χρόνου. Προτάσεις λοιπόν υποστήριξης ε, αυτής της ενεργού ένταξη με δημιουργία θέσεων απασχόληση, με συγκεκριμένα δικαιώματα ε, σχεδιασμένων ειδικά για τις γυναίκες, για τους ανέργους, γιατί μεταξύ των ανέργων ε, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι γυναίκες σε κάποιες χώρες, όπως στην Πορτογαλία. Επίσης, ε, πώς θα υποστηρίξετε τις ε, γυναίκες που, έχουν, που λαμβάνουν πολύ χαμηλές συντάξεις. Στην χώρα μου, παραδείγματο χάρη, ένα σημαντικό ποσοστό των ηλικιωμένων γυναικών παίρνουν ε, σύνταξη 300 ευρώ ή ακόμη και λιγότερο από 300 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνετε ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν, σε τι κατάσταση φτώχειας ζουν εκατομμύρια ε, γυναίκες, εκατομμύρια άνθρωποι. Επίσης, χρειαζόμαστε όντως καλύτερες υπηρεσίες ε, κοινωνικής ασφάλισης και ε, καλύτερες υπηρεσίες του τομέα της ε, υγείας. Εξού και η οδηγία για τα θέματα υγείας. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, θα μπορούσατε να μας πείτε τι προτίθεται να κάνει η Προεδρία. Ε, ευχαριστώ. Ε, ε, ίσως ε, θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στην Υπουργό να απαντήσει <clears throat> και μετά προχωρούμε στον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Ευχαριστούμε. Ήταν πολύ καλές οι ερωτήσεις σας. Θα αρχίσω με τις ερωτήσεις Ελίζα Μπεθλίν. Πρώτον, η οδηγία για την κατάρχηση της διακριτικής μεταχείρισης δεν είναι στο δικό μου χαρτοφυλάκιο, αλλά όταν έρθει ο αρμόδιος υπουργός μπορείτε να την ξαναθέσετε την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα και φυσικά πρέπει να ε, εγκριθεί, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ ε, είναι δουλειά του αρμόδιου Υπουργού. Τώρα, για το θέμα των ηλικιωμένων και για τις βέλτιστες ε, πρακτικές. Πιστεύω, είμαι πεπισμένη ότι τα κράτη-μέλη έχουν έχουν πάρα πολλά να μάθουν το ένα από το άλλο με την ανταλλαγή των εμπειριών, αλλά πρέπει επίσης να βρούμε τρόπους να κάνουμε benchmarking, συγκριτική αξιολόγηση και να χρησιμοποιήσουμε τα καλύτερα παραδείγματα από κάθε χώρα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλω το ζήτημα των ηλικιωμένων να εγγραφεί πιο μόνιμα στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να έχουμε μια πιο διαρθρωμένη ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών και συγκριτική αξιολόγηση ανάμεσα στις επιδόσεις των κρατών μελών. Γι' αυτό σας μίλησα για την μέθοδο του ανοιχτού συντονισμού, για να μάθουμε ένας από τον άλλον. Το χρειαζόμαστε, γιατί η πρόκληση της ε, ε, γύρανσης του πληθυσμού ε, μας αναθέτει ένα πάρα πολύ σημαντικό καθήκον για το μέλλον. Και οι διάφορε πολύ ενδιαφέρουσε προϊούσε εργασίε ε, στα κράτη-μέλη μας επιτρέπουν να, προ... να οδεύσουμε προς αυτή την κοινή πλατφόρμα για να, υπάρχει... να γίνεται σίως αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. Για την αντοχή στα αντιβιωτικά, θα ήθελα να σας πω κάτι, να κάνω κάποια σχολεία, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα. Στα πλαίσια της Επιτροπής Περιβάλλοντος, η Σουηδία ήδη έθεσε το ζήτημα ως προτεραιότητα η συνταγογράφηση των φαρμάκων έχει τόσο κεντρικό ρόλο ε, ε, διότι πρέπει να μειώσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών ούτως ώστε και στο μέλλον να έχουμε ε, αποτελεσματικά, δραστικά αντιβιωτικά όταν πραγματικά τα χρειαζόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα. Επίσης, τονίσαμε ή μάλλον να το θέσω διαφορετικά το ζήτημα. Μαζί με τη Γαλλία και την ε, Τσεχία, στην Τρόικα δηλαδή, συζητήσαμε το θέμα και εμείς από πλευράς μας ε, εστιάσαμε την προσοχή μας στο εξής ε, που δεν έχουμε προαναφέρει. Πώς μπορούμε να ε, βρούμε νέα κίνητρα για τη φαρμακοβιομηχανία για να αναπτύξει νέα αντιβιωτικά, γιατί χρειαζόμαστε νέα προϊόντα, νέα φάρμακα στην αγορά, γιατί τα παλιά δεν πρόκειται πλέον στο μέλλον να είναι δραστικά και αποτελεσματικά. Τώρα, σε σχέση με τις ερωτήσεις Σίλτα Φιγκυρέντη. Η επιπτώσεις οικονομικής κρίσης. Ε, γι' αυτό μας μιλήσατε και πώς επηρεάζει την κατάσταση στον κοινωνικό τομέα. Από Σουηδική Σκοπιάς μας απασχολεί πάρα πολύ η υψηλή ανεργία των ανέργων, ε, των νέων ανέργων, που δεν έχουν να πάνε στη δουλειά το πρωί. Ε, είναι δύσκολη αυτή η κατάσταση. Ε, όταν έχει βρεθεί κάνει σε αυτή την κατάσταση να επανέλθει τελικά στην αγορά εργασία. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα. Ε, στη χώρα μας ε, δεν ισχύει αυτό που είπατε ότι είναι πιο εκτεθειμένες οι γυναίκες από τους άντρες, αλλά αυτό δεν ισχύει σε όλες τις χώρες. Και όντω ε, πρέπει να τονίσουμε ότι είναι μάλλον εθνική αρμοδιότητα αυτό το θέμα, γιατί είναι τόσο διαφορετικέ οι καταστάσει. Αλλά υπάρχουν και κοινά σημεία συγκεκριμένα ότι αυτοί ε, που σε περίοδο οικονομική ύφεση αποκλειστούν από την αγορά εργασία μπορεί να χρειαστούν πάρα, πάρα πολύ, πολύ χρόνο για να επανέλθουν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε νέε θέσει απασχόληση και πρέπει να φροντίσουμε τόσο ώστε ε, κατά τη διάρκεια τη οικονομική κρίση να μπορούν να διατηρούν τι θέσει του, ε, τι θέσει απασχόληση οι άνθρωποι. Τώρα μπορεί να διαφοροποιούνται τα κράτη-μέλη ανάλογα με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, αλλά πάντω ε, ένα σημαντικό στόχο να διατηρήσει κανεί τη θέση του τη δουλειά του. Ε, και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με την ανταλλαγή εμπειριών, με τα καλά παραδείγματα. Όσοι δηλαδή επιτόπου έχουν χρησιμοποιήσει, όπως απέδειξε η πράξη, ε, αποτελεσματικά εργαλεία, μπορούν να τα μοιραστούν με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Μπορούμε να μάθουμε μένα από τους ΔΕ για τον προπολογισμό τώρα. Ε, ουσιαστικά δεν μπορώ να το σχολιάσω το θέμα σε μεγάλο βαθμό. Μπορώ να σας μιλήσω όμως για τον εθνικό μας προϋπολογισμό, δηλαδή πώς δίνουμε προτεραιότητα στις ενεργείς ε, λύσεις στον τομέα της απασχόλησης για το, στον τομέα των γενικών καθολικών υπηρεσιών κοινή ωφέλεια, ε, στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η κρίση να μην πλήξει τα τους πλέον ευάλωτους ε, συμπολίτες μας για τον κοινό προϋπολογισμό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις επιπτώσεις της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης ε, όταν καταρτίζουμε τον κοινό προϋπολογισμό. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Έχουμε ένα τέταρτο ακόμη στη διάθεσή μας και έχουμε πέντε ομιλητές. Κλείνω τώρα τον κατάλογο των ομιλητών και σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε σύντομοι. Μην αρχίσουμε τώρα με την υπέρβαση του χρόνου ομιλίας ήδη από τώρα. Ο κύριος Σέρκας και η κυρία Σιλβάνα Ράπτη συνέχεια. Ο κύριος Σέρκας πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και την κυρία Υπουργό. Ε, πολύ σύντομα θα ήθελα να σας κάνω ένα σχόλιο και να σας θέσω και μία ερώτηση. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι αναφερθήκατε ε, με πολύ καλό τρόπο στα θέματα της τρίτης ηλικίας, στα θέματα του κοινωνικού αποκλεισμού και της ένδυας. Το σχόλιο μου, κυρία Υπουργέ, είναι ότι ούτως ή άλλως κάθε έξι μήνες έρχεται ε, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου ε, και μας κάνει μια διάγωση της κατάστασης. Η κατάσταση είναι ανησυχητική, η διάγνωση είναι πάντα ανησυχητική, αλλά δεν έχουμε ποτέ θεραπεία. Και εμείς ως ε, Ευρωπαίοι θέλουμε όχι μόνο ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες να μαθαίνουν τη διάγνωση, αλλά να τους δίνουμε και μια θεραπεία για την κατάσταση. Και φαίνεται ότι ο ανοιχτός ε, συντονισμός και η μέθοδος ανοιχτού συντονισμού ε, είναι μεν ε, σημαντική, αλλά δεν είναι επαρκής. Ε, αν δούμε το θέμα της ένδυας, όπως είπατε και εσείς, θα έχουμε και το έτος στόχος του χρόνου. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πιο συγκεκριμένα μέτρα. Δεν ξέρω αν θα το κάνετε στη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας ή στη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας. Ε, θα εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι θα έχουμε τον παγκόσμιο έτος κατά της έμβειας για να κάνετε κάτι για την φτώχεια. Ε, το Κοινοβούλιο ανησυχεί ιδιαίτερα για το θέμα της συνέχεια της οδηγίας για, τις, για τη διαμεθοριακή ε, περίθαλψη. Ε, καθυστέρησε, είναι στο Συμβούλιο. Τι γίνεται όμως με την οδηγία αυτή στο Συμβούλιο. Και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω τη Σουηδική ε, Προεδρία αν είναι σε θέση, δεδομένου ότι οι απόψεις εδώ στο Κοινοβούλιο ερίζουν ε, και αν τεθεί το θέμα σε δεύτερη ανάγνωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι αμφισβολίες που έχουμε για το διπλό, διπλή νομική βάση και για οτιδήποτε άλλο. Ε, ξέρετε λοιπόν ότι δεν είναι εύκολη κατάσταση στο Κοινοβούλιο. Εσείς τη γνωρίζετε, είστε διατεθειμένοι να βοηθήσετε και να οδηγήσουμε σε συνένεση. Κυρία Σιλβάνη Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Να καλωσορίσω την κυρία Υπουργό, να την ευχαριστήσω για την ενημέρωση που μας έκανε και να πάρω αφορμή από ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που ανέφερε, το θέμα του Αλτσχάιμερ και της αξιοπρεπούς του δικαιώματος στην αξιοπρεπή γύρανση. Ε, το θέμα του Αλτσχάιμερ ε, έχει άμεση σχέση και με τη μακροχρόνια μέρημνα και με την μέρημνα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν ρωτώ α, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αν υπάρχουν προγραμματισμένες ενέργειες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών που θα μπορούσαν να ωφελήσουν άλλες χώρες για να οδηγηθούμε σε ένα κοινό σχέδιο δράσης για τα επόμενα πέντε χρόνια σε σχέση με τη μακροχρόνια μέρημνα. Το δεύτερο ερώτημα ε, αφορά την μέρημνα για ασθενείς στο σπίτι. Και αυτό το θέτω γιατί εδώ τίθενται πολλά ζητήματα, εγείρονται πολλά ζητήματα σε σχέση με τα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ αρμοδιοτήτων και ευθυνών ανάμεσα στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Στην πατρίδα μου, στην Ελλάδα, έχουμε τεράστιο πρόβλημα στον ιδιωτικό τομέα. Άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο σπίτι, προσφέρουν μέρημνα, αλλά είτε είναι ασφάλιστοι είτε δεν πληρούν προδιαγραφές και ρωτώ εάν προβλέπετε η καθιέρωση ελάχιστων προδιαγραφών μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για τις ανάλογες αρμοδιότητες, κάτι που εκτιμώ ότι θα βοηθούσε πολύ στην πολιτική αντιμετώπιση και στη θέσπιση ενός εθνικού σχεδίου δράσης, εθνικών σχεδίων δράσης και ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης περαιτέρω. Σας ευχαριστώ. Merci, madame. Και εμείς σας ευχαριστούμε κυρία Αντελή και τον Τόμας Μαν. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Εγώ θα αναφερθώ ε, για την, στην υγεία των νέων. Ε, ε, πολλοί είναι οι λόγοι που πλήττουν αν θέλετε την υγεία των νέων, η κακή δίαιτα αν θέλετε, το ότι δεν έχουν δουλειά κλπ. κλπ. Αλλά κυρίως η πρόσβαση στα νοσοκομεία και στις υπηρεσίες υγείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω, γι' αυτό σας ρωτώ ποιες συγκεκριμένες προτάσεις θα δώσετε, για, θα κάνετε ούτως ώστε να δώσετε ξανά πρόσβαση στους νέους αυτούς ε, μελλοντικά. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τόμας Μάνου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Υπουργό που είναι εδώ και χαίρομαι που μας είπε ότι θα φροντίσει να υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ε, για θέματα υγείας και φροντίδας των ηλικιωμένων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πραγματικά είναι ε, πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε το δράμα που υπάρχει σχετικά με τις φαρμακοβιομηχανίες και είναι πολύ σημαντικό τομέα αυτό. Τυχαίνει να τον ξέρω και όλα λιγάκι. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί είπατε ότι θέλετε ε, να ε, γερνούν αξιοπρεπώς οι άνθρωποι και είπατε ότι από τη μια μεριά υπάρχει, υπάρχουν τα γυροκομεία αν θέλετε τα δημόσια και από την άλλη μεριά υπάρχει η ιδιωτική φροντίδα τι εννοείτε όταν λέτε από τη μια είναι το ένα από την άλλη το άλλο ποιες ε, ε, ε αυτή τη διάκριση που κάνετε μεταξύ των δύο αυτών πραγμάτων θα ήθελα να μου την εξηγήσετε λίγο παραπάνω Πρόεδρος, τελευταία μιλήτρια, κυρία Ελίζα Μπετμογάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρίε Υπουργέ για την παρουσίασή σας την οποία εκτίμησα ιδιαίτερα και η οποία είχε κάποιους ιδιαίτερα ανθρώπινους τόνους σε σχέση με τη φροντίδα των ηλικιωμένων και με την αξιοπρεπή γύρανση. Εγώ θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας και να σας ρωτήσω τι φροντίσετε, τι έχετε σκοπό να κάνετε σε αυτούς που φροντίζουν τους ηλικιωμένους, τους φροντιστές ας το πούμε των ηλικιωμένων ε? γιατί ειλικρινά όταν υπάρχουν δύο αν θέλετε όταν ένα, το ζευγάρι στο ζευγάρι υπάρχουν δύο άτομα ο ένας φροντίζει τον άλλον κάποια στιγμή τα πράγματα αλλάζουν ε, κάποιος πάει στο νοσοκομείο ο άλλος μένει μόνο τέλος πάντων ε, πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να βοηθηθούν από, το, από τις συλλογικέ δομές στον τομέα υγείας. Σας ευχαριστώ για τη θέσμευση που δείχνετε και για τις ερωτήσεις σας. Θα αρχίσω με τον κύριο Σέρκας για την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού που έδειξε ότι δεν επαρκεί, όπως μας λέει ο κύριος Σέρκας. Ναι, ναι, συμφωνώ. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτός ο τομέας είναι τομέας εθνικής αρμοδιότητας, ε, κατά κύριο λόγο. Αλλά μπορούμε να υποφεληθούμε από τις εμπειρίες ε, των άλλων κρατών μελών και αυτή η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού θα ενισχυθεί περί ε, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί μαζί μας για άλλα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν το φθινόπωρο. Ήδη λειτουργεί ουσιαστικά αυτή η ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, αλλά θα βελτιωθεί. Πάντω υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Να δούμε πώ μπορούμε να τη, συγγνώμη, να τη διαμορφώσουμε για να λειτουργεί ακόμη καλύτερα. Μπορούμε να το καταφέρουμε μαζί για την διασυνοριακή περίθαλψη τώρα. Δεν είναι θέμα του χαρτοφυλάκιου μου. Ο Γέραν Χέγκλουντ, ο συνάδελφό μου, είναι αρμόδιος. Αλλά τέλος πάντων, να σας εξηγήσω ότι η φιλοδοξία μας είναι να εγκριθούν αποτελε... Ε, συμπεράσματα του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο έχει εργαστεί πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Το γνωρίζουμε. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα σε επίπεδο Συμβουλίου. Εν πάση περιπτώσει, εμά ο απότερο στόχο μα είναι φέτο το Δεκέμβρη να εγκριθούν συμπεράσματα στο Συμβούλιο. Ε, ελπίζουμε ότι θα έχουμε υποστήριξη από τα λοιπά, ε, λοιπά κράτη-μέλη. Ελπίζουμε να θεωρήσουν ότι είναι καλή η πρόταση που θα υποβάλουμε. Τώρα, το θεματικό έτος, το 2010, για τα θέματα της στόχιας, είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, διότι ε, χάρη σε αυτό, κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας, εμείς μπορούμε να προετοιμάσουμε τη βάση, αν θέλετε, για το, αυτό το έτος το 2010. Θα αναλάβει τη σκητάλη η Ισπανική Προεδρία και θα διοργανώσει διάσκεψη για αυτό το ζήτημα σύντομα μετά την ανάληψη της Προεδρίας. Και γι' αυτό κάνουμε και εμεί τη διάσκεψη, αυτή την 8η διάσκεψη Τράπεζα. τράπεζας. Ε, θεωρούμε ότι θα είναι πολύ σημαντικό input, πολύ σημαντική συνεισφορά για την εισαγωγή αυτής τη θεματική χρόνια. Αλλά φυσικά ενεργά πρέπει να εργαστούν και τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο. Για την κυρία Σιλβάνα Ράπτη τώρα. Μου μιλήσατε για το Αλτσχάιμερ. Και το βάρος και τη σημασία της φροντίδας στο σπίτι. Μπορώ πάντα να συμφωνήσω μαζί σας και θα ήθελα να τονίσω ότι ε, πρέπει να βρούμε καλά παραδείγματα σε κοινωνίες που λειτουργούν αισίως και στη διάσκεψη των εμπειρογνωμών εμείς θα μας τα παρουσιάσουμε αυτά τα παραδείγματα, αυτές τις πρακτικές είναι η διάσκεψη που θα γίνει στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου που σας είπα ε, γιατί θέλουμε να βασιστούμε σε αυτά τα καλά παραδείγματα, στις καλές πρακτικές για να διαδοθούν στην Ευρώπη και στην διάσκεψη εμπειρογνωμόνων. Άλλο στόχος είναι να καταλήξουμε σε κρατεά συμπεράσματα στα οποία θα βασιστούμε για να εργαστούμε περαιτέρω και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως ε, βάση για να εγγραφεί πιο μόνιμα το θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ένωσης για τις ελάχιστες ε, ε, απαιτήσει τώρα για την κοινωνική ασφάλιση για όσους ε, φροντίζουν ηλικιωμένους στον ιδιωτικό τομέα. Ε, δεν είχαμε πρόθεση να το γύρουμε αυτό το ζήτημα, να το εξετάσουμε, γιατί είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας και ω εκ τούτου δεν προτιθέμεθα να το εξετάσουμε αυτό το θέμα. Ε, κατόπιν, η υγεία των νέων. Ακούστηκε μία ερώτηση υπάρχουν πάρα πολλές ε, προκλήσεις για την υγεία των νέων. Έχουμε το πάχος, την παχυσαρκία, ε, την προληπτική εργασία που πρέπει να γίνει, το αλκοόλ, παραδείγματος χάρη κατάχρηση του αλκοόλ ε, είναι προτεραιότητα για μας. Θα γίνει διάσκεψη εμπειρογνωμών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και αυτά το Σεπτέμβριο θα γίνουν. όλα αυτά πρέπει να δείτε ότι είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, ε, να διαμορφώσουμε τη συμπεριφορά των νέων, να τους υποστηρίξουμε ε, και κατά τη διάρκεια της Προεδρία μας ο στόχος μας είναι να επιτεθούμε στα διάφορα προβλήματα από πολλές και διαφορετικές ε, πλευρές. Στη συνέχεια, ερώτηση του κυρίου Μαν. που ήθελε να μία διευκρίνηση. Δηλαδή τι εννοούμε να εστιάσουμε στις ατομικές ανάγκες. Να σας εξηγήσω. Είναι κεντρική σημασία. Πρέπει η εστίαση να φύγει από μια γενική περίθαλψη των ηλικιωμένων και να ε, κατευθυνθεί προς τις ατομικές ανάγκες των ηλικιωμένων. Δηλαδή να ε, δημιουργήσουμε ένα σύστημα περίθαλψης ε, το οποίο όμως θα ταιριάζει σε κάθε έναν από αυτούς τους ηλικιωμένους. Και αυτό δεν συμβαίνει συνήθω ότι τα κοιτάζουμε και προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τα συστήματα από την ατομική σκοπιά. Μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί άλλα κριτήρια και γνώμονε. Τι είναι καλό για το προσωπικό, παραδείγματο χάρη. Ή ε, δομές ε, εγκατεστημένες που όμω δεν ταιριάζουν καθόλου στους ηλικιωμένου γιατί δεν μοιάζουν όλοι οι ηλικιωμένοι. Ε, είναι άτομα μοναδικά. Κάθε ένα ηλικιωμένο είναι ένα μοναδικό άτομο όπω ακριβώ και όταν ήταν νέο. Και άρα ε, χρειαζόμαστε μία περίθαλψη των ηλικιωμένων που να λαμβάνει υπόψη τις ατομικές ανάγκες του κάθε ηλικιωμένου. Αυτό έχει ζωτική σημασία. Ε, Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε τη σκοπιά υπό την οποία εξετάζουμε το σύστημα της περίθαλψης των ηλικιωμένων. Αυτό είναι μια βασική αποστολή που θέλουμε να επιτελέσουμε. Μια μεγάλη φιλοδοξία που έχουμε για την ε, Σουηδική Προεδρία να αλλάξουμε την οπτική γωνία. Να, τα, να το δούμε μέσα από το πρίσμα του ίδιου ηλικιωμένου. Για τα παραποιημένα και ψευδεπίγραφα φάρμακα θα ήθελα να σα παραπέμψω στον Γιώραν Χέγκλουντ γιατί ασχολείται επισταμένα με αυτά τα ζητήματα. Οπότε οπότε μπορεί εκείνος να σχολιάσει καλύτερα τα σχετικά θέματα. Η κυρία Μογά μας μίλησε για τη σημασία των ε, συγγενών ε, στην ε, περίθαλψη των ηλικιωμένων, γιατί ασχολείται 24 ώρες το 24, 365 μέρες το χρόνο με τους ηλικιωμένου. και πρέπει κάποιος επιτέλους να λάβει υπόψη και τις δικές τους ανάγκες. Και ξέρουμε όλοι ότι θα καταρρεύσει το σύστημα περίθαλψης αν απεργήσουν ε, οι συγγενείς, αν ε, πετάξουν την πετσέτα και να πούνε λοιπόν όχι, εγκαταλείπω, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πρέπει να του υποστηρίξουμε ε, για να επιτελέσουν τα καθήκοντά του. Με διάφορου τρόπου στη Σουηδία, παραδείγματο χάρη, τροποποιήσαμε την νομοθεσία μα και είπαμε ότι δικαιούνται και εκείνοι παροχέ για να εξεταστούν και οι δικέ του ανάγκε. Να κι άλλος ένας λόγος για την ανταλλαγή των εμπειριών στα θέματα των ηλικιωμένων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ε, φυσικά ε, μιλάμε για τους συγγενείς των ηλικιωμένων, ε, τα κοντινά τους πρόσωπα, ε, που πρέπει να κερδίσουν το χρυσό για τις προσπάθειες που κάνουν και σπάνια κανείς τους ευχαριστεί. Πάντως εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς για τις ερωτήσεις σας. Καλή επιτυχία με τη νέα θητεία και τους προσεχείς μήνες, τους φθινοπορεινούς. Ελπίζω να έχουμε αγαστή συνεργασία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τις σαφείς απαντήσεις σας ε, στα ερωτήματα που ετέθησαν. Ξέρουμε ότι έχετε που υποχρεώσεις και αλλού τι να κάνουμε. Αυτό είναι το καθήκον των διαφόρων υπουργών που προεδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε στο μέλλον. Καλό κουράγιο και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Ξαναγυρνώ βέβαια στο σημείο 1, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο 7 δεν θα το συζητήσουμε σήμερα όπως είπα και πιο πριν και δεν πρόκειται αύριο να ψηφίσουμε το σημείο 12 κατά συνέπεια. Επίσης δεν θα ψηφίσουμε και για το αφού δεν θα έχουμε συζητήσει το θέμα και θα συζητήσουμε και για τη γνωμοδότηση για τις γυναίκες από την Επιτροπή Γυναικών θα το δούμε το θέμα αυτό αργότερα τώρα ε, για τα πρακτικά της συνεδρίας 16 Ιουλίου αυτά πρέπει να τα εγκρίνουμε ε, μέχρι το τέλος της συνεδρίας πείτε μου αν έχετε πρόβλημα ε, τώρα για το για το τις ανακοινώσεις της Πρόεδρου να σας πω δυο λόγια για το web streaming δηλαδή όλες οι συζητήσεις μας περνάνε κατευθείαν στο ίντερνετ στο διαδίκτυο και μπορούν να τις παρακολουθήσουν όλοι παντού ε, κατά τα άλλα Υπάρχουν δύο ανακοινώσεις, μια για την διαδικασία του προπολογισμού 2010 και άλλη μία και ε, το, για τον προπολογισμό 2010 τμήμα 3 επιτροπή το έχουμε το θέμα και στη μερισή διάταξη πρέπει να υπάρχεται ο κύριος Σερκάς Κυρία Πρόεδρε λυπούμε πάρα πολύ που σας διακόπτω αλλά ε, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να μου εξηγήσετε εάν ε, σήμερα κάνουμε κάποιες αλλαγές σχετικά με τις αποφάσεις που πήραν τον Ιούλιο οι συντονιστές. Συγγνώμη, ε, ε όταν ε, δεν ψηφίζουμε για κάποια έκθεση ενώ έχει κανονιστεί ψηφοφορία πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος διαφορετικά δεν είναι δημοκρατική κατάσταση συμφωνώ ε, γιατί να μην γίνει η ψηφοφορία. Ε, το συζήτησα το θέμα με την Πρόεδρο. Η Επιτροπή και τα συνδικάτα προσπαθούν να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Τα δύο μέρη δήλωσαν ότι χρειάζονται και άλλο χρόνο. Θα έπρεπε ίσως λοιπόν να δεχτούμε την πρόταση της Προέδρου. Όμως ε, για την τελική απόφαση δεν γνωρίζω ποια θα είναι η καλύτερη λύση γιατί είναι κανθώδες το ζήτημα. Νομίζω στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών καλό θα ήταν να συζητηθεί το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Αν κατάλαβα καλά και οι δύο παρεμβάσεις αναφέρουν το σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης για το χρόνο εργασίας ε, αυτών που ασχολούνται στις οδικές μεταφορές. Δεν ξέρω αν η συγγήτρια, η κυρία Edith Bauer θέλει να κάνουμε την ανταλλαγή απόψεων. Εγώ δεν βλέπω γιατί να την κάνουμε όταν η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν είναι παρόντα διότι δεν εκκλήσισαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ κυρία εισηγήτρια προτείνω να ακολουθήσουμε τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αν μετά τη συζήτηση του σημείου 5 για τον προϋπολογισμό ε, έχουν έρθει ή μπορούν να έρθουν εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου τότε να τα, το συζητήσουμε το θέμα σας. Τι να σας πω κύριος Τούσας. Ναι κύριε Πρόεδρο, ε, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να αναφερθώ σε ό,τι αφορά την ε, ημερήσια διάταξη. Ο καθορισμό τη ημερήσια διάταξη δεν έχει ένα τυπικό χαρακτήρα και η έναρξη των εργασιών και τη εξέταση των θεμάτων από την Επιτροπή απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων. Έχει ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο και ουσία και προσδιορίζεται με βάση τον κανονισμό και τις αποφάσεις των μελών της Επιτροπής μας. Αν λοιπόν κάτι πρέπει να αλλάξει, σε προγραμματισμένες αποφάσεις, στη διαμόρφωση, θα πρέπει να ακολουθούν αυτές οι διαδικασίες. Έτσι το ότι δεν παρευρίσκεται σήμερα εκπρόσωποι από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο, δεν ξέρω ποιος πήρε αυτή την πρωτοβουλία να μην τους καλέσει. Και έχει τέλος ε, πάντων ε, ευθύνη. Κύριε Τούσα, ένα λεπτό επιτρέψτε μου να πω ορισμένα πράγματα. Η κανονική ημερήσια διάταξη που εγκρίθηκε ε, και ενημερώθηκαν σχετικά και η Κομισιόν και το Συμβουλίο, οι εκπρόσωποι της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Η ημερήσια διάταξη λοιπόν που εγκρίθηκε έλεγε στο σημείο 6 ε, το, ε, το θέμα από την Επιτροπή των γυναικών και παρακάτω οργάνωση του χρόνου εργασίας των γυναικών που εκτελούν ε, τις ε, κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Μετά τι έγινε. Η κυρία Edith Μπάουερ θέλει τώρα να αντιστραφούν τα σημεία 6 και 7 της ημερήσιας διάταξης. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το σημείο 7 πριν από το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Αν, αν τελικά μπορέσουμε να, τους, να πούμε στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο να έρθει πιο μπροστά να έρθουν πιο πριν. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κανένα θέμα περαιτέρω. Ξεκινούμε αμέσως με το σημείο 5 της σημερινής διάταξης και εντωμεταξύ μέχρι να τελειώσουμε το σημείο 5 του προπολογισμού θα δούμε αν μπορούμε να συζητήσουμε αμέσως μετά το σημείο 7. Για το 5 Προϋπολογισμός 2010. Ο εισηγητής είναι ο συνάδελφός μας Λάζλος Ζιουζάν. Ε, ε, ε, Κύριε Ωρί, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Σουρζάν είναι ε, ο εισηγητής από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εγώ είμαι ο εισηγητής αυτής εδώ της Επιτροπής. Ζητώ συγγνώμη, λέει πρόεδρος. Παρακαλώ. Ωραία, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος ξεκινήσαμε τη δουλειά μας ήδη από την περασμένη θητεία ε, για το προπολογισμό του 2010 ε, έγιναν πολλές ε, ε συζητήσεις ε, και εδώ και αλλού και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η σε τελευταία ανάλυση η Επιτροπή Προπολογισμών θα εγκρίνει το προπολογισμό. Εμείς απλώς ε, ιεραρχούμε κάποιες προτεραιότητες, προτείνουμε κάποιες προτεραιότητες, κάποια συγκεκριμένα πράγματα για συγκεκριμένα κονδύλια. Η Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως στην κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού μάλλον του πρόσχεδιου προπολογισμού ε, δεν έλαβε υπόψη και πολύ σημαντική και, και πολύ τις κοινοβουλευτικές επιτροπές οφείλουμε να πούμε αυτή είναι εν πάση περιπτώσει η εμπειρία μας από το παρελθόν ωστόσο εδώ βλέπω ότι πολλά από τα πράγματα που ε, είπαμε ε, θα πρέπει να ε, τα επαναλάβουμε όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτική γιατί δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν τα παιδάκια που πάνε στο παιχνιδάδικο με τους γονείς τους και επιμένουν να τους πάρουν οι γονείς όλα τα παιχνίδια που τυχαίνει να τους αρέσουν. Λοιπόν, εδώ όντως έχουμε κάνει πολλές προτάσεις και εγώ πάρα πολλές τροπολογίες υπέβαλα ε, αλλά υπάρχουν και πολλές τροπολογίες άλλων ε, συναδέλφων τις οποίες προσπάθησα να ε, ε, ενσωματώσω στην έκθεσή μου. Έχετε μπροστά σας φαντάζομαι τις τροπολογίες. Ρίξτε μια ματιά στο κείμενο. Παράγραφη Δύο, 3, εγώ είμαι υπέρ, τέσσερα είμαι υπέρ, πέντε, τροπολογία της κυρίας Φεγκρέιντο είμαι υπέρ, το έξι, την έξι όχι, Γκέντς. ναι, 8 είναι η τροπολογία Γκέντς. Εκεί έχω κάποιο πρόβλημα, το ίδιο και με την εννιά του κυρίου Χιούζ. Ε, που σχετίζονται με το θέμα των μικροπιστώσεων. Η κυρία Γκέντς λέει ότι ο κύριος Χιούς λέει ότι όταν συζητήσουμε τα μικροκονδύλια, τα μικροδάνεια, τότε θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε ορισμένα πράγματα. Κυρία Γκόνιτς, έχετε την αντίθετη άποψη. Είναι αντιφατικές λοιπόν οι δύο αυτές τροπολογίες 8 και 9 ο, η 8 λέει τέρμα η συζήτηση ή προδικάζουμε τη συζήτηση με μια έννοια αν θέλετε και αυτό, αυτή την τροπολογία εγώ δεν μπορώ να αντιδεχτώ τη, η 9 είναι πολύ πιο ανοιχτή η τροπολογία και θα μπορούσα να τη δεχτώ το, η, το, η 10 αναφέρεται σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα είμαι υπέρ είμαι βρίσκει σύμφωνο η ιδέα, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπευλήθη, ε, υποβάλλεται εδώ λίγο αργά. Όταν πρωτεία προγράμματα πυλ ε, υπάρχει μια περιορισμένη χρηματοδότηση για ορισμένα, για τέσσερα παραδείγματο χάρη. Από εκεί και πέρα, άμα προχωρήσουμε παραπάνω και φτάσουμε στα 6, 7 και τα λοιπά, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι δεν είναι ρεαλιστικό να δεχθούμε την τροπολογία αυτή εδώ σήμερα. Είναι μάλλον αργά. Τώρα δεν θα σας ε, ενοχλήσω αναφέροντας συγκεκριμένε θέσεις ε, του προϋπολογισμού, ε, γύρω στις 50 τροπολογίες έχουν υποβληθεί. Ε, γενικά λέω ότι οι σοσιαλιστές ζητούν ζητούν χρηματοδότηση για τα αυξημένη για το progress 500 εκατομμύρια επίσης θα ήθελα να είναι δυνατόν το, για, το, για τα μικροδάνεια, μικροπιστώσεις δεν μπορούμε. Το Συμβουλίο έχει βάλει ένα συγκεκριμένο ποσό. Ε, ε, νομίζω ότι είναι, δεν είναι σκόπιμο να μιλούμε για συγκεκριμένα ποσά εδώ τα οποία να ζητούμε. Μια συμβαστική λύση κατά την άποψή μου θα ήταν να έχουμε μία ειδική θέση στον προπολογισμό όπως προτείνουν οι σοσιαλιστές η οποία όμως να μην περιλαμβάνει νούμερο ε να λέμε πρόσημο και να βάλουμε το νούμερο αργότερα. Επίσης έχουμε το πιλωτικό σχέδιο σχετικά με ταυτιστικά άτομα. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ιδέα, αλλά φοβούμαι ότι είναι πολύ αργά για να ζητήσουμε χρηματοδότηση και για αυτό το πολιτικό πρόγραμμα. Ας δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να περάσουν έξι προγράμματα πιλωτικά. Ε. Δίκιο είναι καλή ιδέα αυτή νομίζω ότι μπορούμε όμως να το ξανά αργότερα το πολιτικό αυτό πρόγραμμα. Αυτά λοιπόν ε, δεν έχω άλλο να συμπληρώσω στην εισαγωγή μου. Περιμένω τα δικά σας σχόλια και ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Ναι, αλλά θα πρέπει ε, να ε, να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και να, να δούμε τα θέματα πάρα πολύ γρήγορα γιατί αύριο πρέπει να ψηφίσουμε αν θέλουμε να πάει το θέμα παραπέρα και να ληφθούμε υπόψη. E, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις ε, για την παρέμβαση του συναδέλφου Όρη. Υπάρχουν ε, κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες για την ε, πρόταση για την μικροχρηματοδότηση. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε μια φάση στην οποία θα μπορούμε να δώσουμε τη συνένεσέ μας σε κάτι τέτοια για να μπορούμε να αποφασίζουμε και κονδύλια στον προϋπολογισμό. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόταση που κάνατε θα μπορούσε να υπάρχει μια γραμμή προπολογισμού ad hoc ξεχωριστή για να μην παίρνουμε τα κονδύλια από τα πιλωτικά προγράμματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αύριο να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε μέσω της ψηφοφορίας για τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για ένα κονδύλιο το οποίο θα ε, προκύψει από άλλα κονδύλια, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, και από άλλες συνεισφορές. Θα μπορούσαμε να κάνουμε λοιπόν μια προφορική τροπολογία για το θέμα αυτό και να συμπεριλάβουμε την πρόταση αυτή. Ένα άλλο θέμα το οποίο έθιξε ο κύριος Σέρι ε, αφορά το θέμα των ε, οδηγών αυτοκινήτου, των, των αυτοκινητιστών οι οποίοι περιλαμβάνονται στο πιλωτικό πρόγραμμα. Οι δυνατότητες που έχουμε είναι περιορισμένες διότι, όπω είπε και ο ίδιο, μπορούμε να υποστηρίξουμε μόνο περιορισμένο αριθμό πιλωτικών προγραμμάτων. Χαίρομαι που ο κύριο Σόρι στηρίζει τουλάχιστον ε, για λόγους αρχής την πρόταση αυτή. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να τον ευχαριστήσω. Euh, Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Βισένσο Γιωβίν από τους Φιλελευθέρους και Νίλαν Κάμπροτ στη συνέχεια. Βισένσο Γιωβίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. για την ε, γνωμοδότηση του κυρίου Όρη ε, είμαι σύμφωνος. Ε, θα πρέπει να την υπερψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Τώρα, για τα όσα προτείνονται στην αρμόδια Επιτροπή για το θέματα προϋπολογισμού επί της ουσίας, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών και δεδομένου ότι θα έχουμε το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ε, ε, και ε, υπάρχει και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μειώσουμε τις παροχές κατά 9% σε σχέση με το 2009. Επίσης θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την επαγγελματική ισοτιμία, κάποια θέματα τα οποία προβλέπουν μια σημαντική αύξηση των κοινωνικών πτυχών και του ενηλοποίηση του προγράμματος πρόγρας. Οι τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής, ο κύριος Όρη, οι 2, οι 3 και οι 12, είναι συνεπακόλουθε αυτών που σας είπα, γι' αυτό και θα πρέπει να τις υπερψηφίσουμε εμείς ως Επιτροπή. Το ίδιο ισχύει και για την ε, τροπολογία υπαριθμών 8, την οποία παρουσίασε η κυρία Γκόσ, ζητώ συγγνώμη για τον τρόπο που προφέρω το όνομα, και η τροπολογία 11 και των κυρίων Γκόσ και Ούνς. Αυτή η τελευταία είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι αφορά την ένταξη στον εργασιοκό χώρο των ε, ατόμων που ε, έχουν αυτισμό. Ε, η πολιτική μου ομάδα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τέτοια πράγματα και είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη. Τώρα, για τη γενικότερη θέση προπολογισμού, σε γενικέ γραμμέ συμφωνούμε με τι αλλαγέ που προτείνει ο εισηγητή, αλλά Όσον αφορά τις τροπολογίες 6317, 6320, 6321 και 6322 που παρουσίασε ε, η ομάδα των σοσιαλιστών, και αφορούν ε, το πρόγραμμα Progress, ε, το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ομάδα των φιλελευθέρων. Σε γενικές γραμμές είμαστε υπέρ. Ε, αλλά θα πρέπει βέβαια να δούμε κατά πόσον καλύπτονται από οικονομικής πλευράς αυτά και κατά πόσον ε, συμφωνεί και ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα εν συντομία να σας παρουσιάσω μία προφορική τροπολογία στο 310243. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης προσαρμογής ε, παγκοσμιοποίησης. Είχαμε 15 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το οικονομικό έτος, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι το ποσοστό ε, εκταμίευσης ήταν πάρα πολύ χαμηλό έχουμε μια εκταμίευση της τάξης του 10%. Μιλάμε δηλαδή ε, για πολύ μικρό ποσό σε σχέση με αυτά τα 15 εκατομμύρια και ουσιαστικά θα μπορούσε κάποιος να δηλώσει ότι είναι άχρηστο αυτό το ταμείο. Θα ήθελαμε λοιπόν ε, να μειωθεί το αποθεματικό, ε, να περάσει στο μισό. Madam Chairman, uh, thank you very much. And, um, Κύριο Σολμερέ, ευχαριστώ Πρόεδρε και απευθύνομαι στους νέους συναδέλφους που ίσως δεν με γνωρίζουν. Ρότζε Χολμε λέγομαι, συντηρητικός από τη Βρετανία και είμαι και ο μόνος εδώ, δεν κάνω λάθος ή μπορεί και να, να, γίνουμε, να ανέβουμε στην κυβέρνηση του χρόνου, οπότε θα εφαρμόσουμε τη δική μας ε, στρατηγική στον τομέα αυτό. και μπορεί και να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά τα ζητήματα. Όλοι θέλουμε εκπαίδευση, όλοι θέλουμε να διατηρηθούν οι θέσει απασχόληση, όλοι θέλουμε να είμαστε καλοί με του αυτιστικού, αλλά υπάρχουν ε, και άλλα άτομα με άλλε αναπηρίε που μπορεί να θεωρήσουν ότι υφίστανται ε, διακριτική μεταχείριση γιατί προστατεύουμε μία μόνο ομάδα ατόμων με αναπηρίες. Πάντως, ε, φανταστείτε τις ε, μπαλίτσε πάνω στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, τι ωραίε που είναι, τα χρώματα κτλ. Έτσι, αυτή την εικόνα έχω με όλα αυτά όπου ακούω, αλλά μην το παραφορτώνετε το χριστουγεννιάτικο δέντρο γιατί θα πέσει κάτω, θα πιάσει και φωτιά το χαλί, τελείωσε έχουμε ποσοστό ανεργία γύρω στα 10%. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στην Επιτροπή. Να ξεκαθαρίσουμε γιατί έχει τόσο υψηλό ποσοστό ανεργίας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει σχέση φυσικά με την παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλά ναι, καθένα και τουλάχιστον τα 10 χρόνια που είμαι εγώ εδώ στο Κοινοβούλιο, ε, οφείλεται επίση ε, ε, στην υπερρύθμιση των αγορών εργασία και ε, στην υπερβολική φορολόγηση και των εταιριών και των ε, ιδιωτών. Ε, δεν είναι ο στόχος να παίρνουμε τα λεφτά από τις ιδιώτες και να τα δίνουμε στους δημόσιους υπαλλήλους που τα δίνουν στα αγαπημένα τους, στα προσφυλή τους προγράμματα. Πρέπει να μειώσουμε τη φορολογία. Ε, τα έχω ξαναπεί αυτά, αυτά και παρόμοια πράγματα. Ξέρω ότι δεν έχω αλλάξει, αλλά επειδή ήρθαν και νέοι συνάδελφοι είπα να τα θυμίσω η κυρία Φιγκυρέιντο και στη συνέχεια η κυρία Λίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις θα κάνω. Πρώτον, για να αιτιολογήσω τις ε, τροπολογίες που υπέβαλα. Ε, ο στόχος είναι να ληφθεί υπόψη η τωρινή κατάσταση με τις ε, σοβαρές επιπτώσεις που έχει στον κοινωνικό τομέα. Να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τους οικονομικούς πόρους, αλλά και να επιστήσουμε την προσοχή σε άλλες ε, πολιτικές που βασίζονται στην υποστήριξη που υπάρχει για τα κοινωνικά ζητήματα και που προάγουν την κοινωνική ένταξη. Παραδείγματο χάρη η προώθηση ποιοτικών κοινοφελών υπηρεσιών, δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος κτλ. Ε, κτλ. Αλλά, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Σιγητά, υπάρχει και ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να μετατραπεί η προσωρινή επισφαλής εργασία σε μια εργασία με πραγματικά δικαιώματα. Αυτό πλήττει κυρίως τους νέους και τις γυναίκες. Σε κάποιες χώρες κάπου γύρω στα 20% της απασχόλησης των ατόμων ε, ή πάνω από 20% ζουν αυτές τις συνθήκες επισφαλούς εργασίας ε, και σχεδόν το σύνολο των νέων θέσεων απασχόλησης είναι τέτοιες θέσεις απασχόλησης. Οπότε πρέπει κάτι να κάνουμε για να δημιουργούνται αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας με δικαιώματα για τους νέους, για τις γυναίκες και για όλους όσους πλήττονται από αυτή την κατάσταση. Επίσης, είναι απαραίτητο για τους ανέργους που δεν επέλεξαν να είναι άνεργοι, έτσι απλά δεν καταφέρουν να βρουν δουλειά. Πρέπει να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς ε, συνθήκες διαβίωσης. Δεν πρέπει να δεχόμαστε να μένουν ε, ξεκρέμαστοι χωρίς καμία κοινωνική στήριξη. και οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης είναι η επιδείνωση της φτώχειας. Ε, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία μας δείχνουν ότι έχουμε πάνω από 22 εκατομμύρια ανέργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι το τέλος του 2009 μπορεί να υπερβεί να υπερβούμε και τους τα 25 εκατομμύρια και να πλησιάσουμε τα 30 εκατομμύρια ανέργους. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε μια τέτοια κατάσταση. Ευχαριστούμε. Διαβάζω τον κατάλογο των ομιλητών. Μπορώ να κλείσω τον κατάλογο και μετά από αυτούς τους τρεις ομιλητές να ακούσουμε την Επιτροπή. Πάρα πολύ ωραία. Η κυρία Λίν. Ευχαριστώ πολύ. Μια διευκρίνηση για ένα θέμα. Στο 6320 από ό,τι ξέρω, οι σοσιαλιστές μπορεί να την αποσύρουν. Ε, δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Ελπίζω όχι, διότι εγώ θα ήθελα να υπάρχει... Ε, μία θέση στον προϋπολογισμό και να αυξάνεται κιόλα για, ε, για τις διακρίσεις. Ε, τώρα, έγινε η παρατήρηση για τον αυτισμό. Υπάρχουν ε, βέβαια και πολλά πιλωτικά προγράμματα για άλλες αναπηρίες. Αλλά το θέμα του αυτισμού ε, είναι πλέον διαπιστωμένο ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων τα οποία έχουν αυτισμό και δεν μπορούν να έχουν θέση εργασία παρά την οδηγία για την απασχόληση. Ήθελα να το διευκρινίσω αυτό, διότι ο αυτισμός είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να υπάρχει μια γραμμή προπολογισμού για το θέμα αυτό κατά την άποψή μου. Η κυρία Τζιν Λάμπερ και μετά η κυρία Μόρα. Κυρία Λάμπερτ, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την ε, μικροχρηματοδότηση. Σαφώς υποστηρίζουμε το άνοιγμα μια γραμμή προπολογισμού για το θέμα αυτό. Επί της αρχής ε, θα είχαμε μεγάλα προβλήματα ε, για να πάρουμε κονδύλια από το Progress, διότι ούτως ή άλλως προσπαθήσαμε τόσο πολύ να βάλουμε χρήματα στο Progress στο παρελθόν. Ε, Μα ικανοποιεί το γεγονό ότι υπάρχει μια θέση στον προπολογισμό γι' αυτό, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε αργότερα πόσα χρήματα ακριβώ θα πάνε εκεί, υπό την προπόθεση ότι θα μα ικανοποιήσει και πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού. Τώρα, για τα πιλωτικά προγράμματα, υποστηρίζουμε την θέση του ε, εισηγητή. Θεωρούμε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να αντιμετωπίσουμε ε, τα επιπλέον πιλωτικά προγράμματα όπως αυτό που προτείνεται για τον αυτισμό. Κατανοούμε ότι υπάρχουν δυσκολίε, αλλά δεν θεωρούμε ότι αυτή, σε αυτή τη φάση αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μόρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 6346 ε, το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ε, Ροσλίν Μπασλό και Ζαν Λουί Κοτινή ήταν αυτοί που έφτιαξαν το ταμείο αυτό δεν είναι πια μαζί μας είναι όμως τέος συναδελφοί μας νομίζω ότι το ταμείο αυτό καταφέραμε να το ε, αναπτύξουμε με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να εξυπηρετεί ε, την, όλο τον κόσμο ε, τους να αναπροσαρμόζει αν θέλετε ή να επιμορφώνει ε, τους εργαζόμενους που δεν έχουν ε, δουλειά ε, και που πρέπει να μάθουν κάτι καινούριο. Νομίζω λοιπόν ότι οπωσδήποτε το ταμείο αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Γι' αυτό είμαι υπέρ της γενικής γραμμής που έχουμε χαράξει και ακολουθούμε εδώ και ε, καιρό σαν Επιτροπή Απασχόληση υπέρ του Ταμείου λοιπόν. Πρόεδρος, η κυρία Ντόνελη, τώρα διευθύντρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα θέλαμε να μας μιλήσετε εσείς τώρα και να επανέλθετε αν είναι δυνατόν στο θέμα αυτό των μικρο δανείων, των μικροπιστώσεων, γιατί είναι ένα αμφιλεγόμενο τελικά θέμα. Και προφανώς, αν θέλετε να αναφερθείτε σε άλλα θέματα, ακόμη καλύτερα. Έχετε το λόγο, κυρία μου. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε και την ε, δυνατότητα να απαντήσω σε κάποιες από τις ε, απόψεις που ακούστηκαν. Για τις μικροπιστώσεις, αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνουμε να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια από το Progress, ε, περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ ε, σε τέσσερα χρόνια, που σημαίνει ότι θα έχουμε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε αυτή την πρόταση να χρησιμοποιούν τα χρήματα από το Progress ως άμεση αντιμετώπιση της κρίσης, διότι θεωρήσαμε ότι αυτοί, αυτές οι μικροπιστώσεις θα επιτρέψουν στα άτομα τα οποία έχασαν τις τέσσερι εργασίας τους ε, λόγω της κρίσης να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας κυρίως ως αυτοαπασχολούμενοι ή ως μικροεπιχειρηματίες. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τηρούμε τις διατάξεις της ε, ε, συμφωνίας, της διοργανικής συμφωνίας και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει κονδύλια από, άλλα, ε, από άλλες θέσεις του προϋπολογισμού, θεωρούμε ότι το progress είναι αυτό το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την περίπτωση. Να κάνω δύο παρατηρήσεις, μία τεχνικής φύσεως. Η αύξηση τη γραμμή προπολογισμού του Progress για να λάβουμε υπόψη και τα κονδύλια τα οποία χρειαζόμαστε για τι μικροπιστώσει, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό ακριβώς την πρότασή μας, η πρότασή μας ήταν ευητή Μία ήταν να κάνουμε μία προσαρμογή του ίδιου του προγράμματο του Progress και η δεύτερη ήταν η δημιουργία μια νέα θέση στον προπολογισμό για να, με τις, να ασχοληθούμε με τι μικροπιστώσει. Από τεχνική σκοπιά, λοιπόν, είναι πολύ πιο εύκολο να έχουμε μια ξεχωριστή γραμμή προπολογισμού παρά να ε, πάρουμε κονδύλια από το Progress, το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να μειωθεί και να επαναδιατεθούν τα κονδύλια. Είναι πολύ περίπλοκο για. Ε, Γι' αυτό ακριβώς ε, ζητήσαμε ε, να έχουμε νέα διάθεση των κονδυλίων για να βελτιώσουμε την κατάσταση σε αυτό. Τώρα, για το Ταμείο Προσαρμογής παγκοσμιοποίηση, ε, σαφώ είναι ένα πολύ σημαντικό ταμείο. Κάθε φορά ανταποκρίνεται όταν υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα. Ε, θα ξέρετε ίσω ότι μόλις τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός ε, και άλλαξε το σημείο 2, τη χρήση του Ταμείου και σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση τη κρίση, φανταζόμαστε ότι το 2010 θα υπάρχουν μεγάλε αιτήσει, μεγάλη ζήτηση για το Ταμείο αυτό. επομένω. δεν θεωρούμε ότι είναι κατάλληλη στιγμή να αλλάξουμε τα ποσά εδώ. Και μια τελευταία παρατήρηση για τα πιλωτικά προγράμματα. Η Επιτροπή πολύ σωστά εντοπίζει ποιε δραστηριότητε καθορίζονται στα πιλωτικά προγράμματα. Να σα επισημάνω όμω ένα πρακτικό θέμα. Το 2010 θα ξεκινήσουμε αυτό το, αυτές τις μικροπιστώσεις, θα έχουμε και το Ταμείο Προσαρμογής ε, της Παγκοσμιοποίησης. Επομένως, ο αριθμός των πολιτικών προγραμμάτων που μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά εκφύσεως ε, θα είναι περιορισμένος. Θα ήταν καλύτερο να μην έχουμε πάρα πολλά. Βέβαια η Επιτροπή σας θα αποφασίσει πόσα θα έχουμε. Βεβαίω η Επιτροπή μας θα μορφώσει άποψη ε, ούτως ή άλλως, αλλά χαιρόμαστε για τα σχόλια που κάνατε. Λοιπόν, ε, κύριε Σιγητά, θέλετε να πάρετε πάλι το λόγο να μας να κλείσουμε τη συζήτηση και να μας υποβάλλετε και συμβαστικές λύσεις ίσως εν ώψη της ψηφοφορίας αύριο. Ναι, πρώτα πρώτα θα ήθελα να απευθυνθώ στην Ελίζαβετ Μόγα η 6346 την οποία ανέφερε ε, είναι ε, πραγματικά ε, ταυτόσιμη με τη μια άλλη τροπολογία, τη μία την υπέβαλα εγώ, ε, οποιαδήποτε από, αυτούς, από αυτές τις δύο μπορούμε να τις διαγράψουμε, είναι ίδιες αλλά κατά τα άλλα μπορούμε να τη δεχτούμε προφανώς. Από εκεί και πέρα. Ε, όσον για την ε, κρίση και την ε, εμπειρία, ε, αν θέλετε, που είχαμε σχετικά με παρόμοια θέματα στο παρελθόν ξέρουμε ε, τι μπορεί ε, να γίνει ήδη από τώρα και με σίγουρο στο μέλλον η για το Ταμείο ε, Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση είναι ακόμη πιο ε, πολλέ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε πράγματα, τα πράγματα όσα έχουν. Ε, προτείνω να διατηρήσουμε τα πράγματα όσα έχουν και γιατί πράγματι το ταμείο αυτό θα μας χρειαστεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Κανείς δεν αμφισβήτησε ε, τε, επί, από τη δουλειά του διαφόρων ιδρυμάτων με τα, τα οποία ασχολούμεθα του Δουβλίνου παραδείγματος χάριν και άλλων που βεβαίως έχουν και αυτά τα ιδρύματα ανάγκη για επιπλέον πόρους. Ε, νομίζω ότι εκείνο που έχουμε να κάνουμε σχετικά, επειδή πρόκειται για πολύ αξιόλογα ιδρύματα, είναι να διατηρήσουμε τα ποσά έτσι όπως τα προτείνει η Κομισιόν. Ωστόσο, πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, ε, είχε τεθεί το θέμα της μείωσης των πόρων που διατίθενται για το πρόγραμμα σχέση με το πρόγραμμα εργασίας η Κομισιόν τότε δεν μας είχε δώσει απάντηση και έκτοτε δεν έχω ακούσει τίποτα σχετικά να ρωτιέμαι περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, Όλα τα ταμεία αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα για την απασχόληση. Θα Πρέπει να αποφύγουμε να γελιοποιηθούμε και να παραμείνουμε ρεαλιστές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζητήσουμε αύξηση αυτή τη στιγμή. Ούτως ή άλλως θα μας αρνηθούν συζήτησα και με τους ε, συναδέλφους από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ε, ξέρω τι γίνεται συνήθως μέχρι τώρα. Ε, επομένως μου φαίνεται ότι η πρόταση των σοσιαλιστών δεν είναι ρεαλιστική. Εξακολουθώ λοιπόν να εμένω στην άποψη ότι πρέπει να περιμένουμε. Πρέπει να περιμένουμε τη συζήτηση για το Ταμείο για τις Μικροπιστώσεις και από εκεί και πέρα θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούσαμε άλλωστε ότι από τεχνική ε, σκοπιά είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστούμε το θέμα δημιουργώντα μια ξεχωριστή ad hoc ε, θέση στον προπολογισμό. Α δημιουργήσουμε λοιπόν αυτή τη θέση στον προπολογισμό και να τη συζητήσουμε του επόμενου μήνε και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει στου επόμενου μήνε. Στη συνέχεια θα αποφασίσουμε τι στρατηγική πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα προκύψει άλλωστε και από την ψηφοφορία λίγο πολύ αυτό. Και ε, έχει δίκιο και η κυρία Γκούνς σε αυτό. Η πρόταση ήρθε έγκαιρα, όχι πολύ καθυστερημένα, αλλά είναι και έξι μήνες πλέον που κάνουμε διαβουλεύσεις, κάνουμε διαπραγματεύσεις για την πρόταση αυτή. Άρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να μιλάμε για την πρόταση αυτή, ε, διότι στο παρελθόν δεν έχουμε συζητήσει τίποτα. Εστιάσαμε λοιπόν σε ένα περιορισμένο αριθμό πολιτικών προγραμμάτων, τα οποία θέλαμε οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν στον προπολογισμό, αλλά εξακολουθώ να επιμένω και εξ ονόματος της ομάδας μου ότι συμφωνώ ε, θα μπορούσαμε κάλλιστα να δούμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα στον επόμενο προπολογισμό. Μάλιστα, θα περάσουμε στην ψηφοφορία αύριο. Όπως σας είπα ε, στην αρχή της συνεδρίασης και για να ευχαριστήσω την κυρία Μπάουερ, ήρθε ε, ο εκπρόσωπος Επιτροπής και το Συμβούλιο μας είπε ότι έχει εμπιστοσύνη στη σοφία του Κοινοβουλίου. Οπότε ας περάσουμε ευθύ αμέσως στο σημείο 7. Τις μερικές διάταξης θα επανεξετάσουμε, ας το πω έτσι, την έκθεση της κυρίας Μπάουερ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, ήθελα απλά να σας πω πως στη συνεδρίαση των συντονιστών που έγινε τον Ιούλιο για, στη συνεδρίαση σύσταση σε σώμα του συντονιστών είχε εγκριθεί αυτή, είχε συμφωνηθεί να παραμείνει έτσι ακέραια χωρίς καμία αλλαγή έκθεση και τα ταχύτερο δυνατό να υποβληθεί στην Ολομέλεια. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ίδιο ο Επίτροπο, για να είμαι συγκεκριμένη, μα κοινοποίησε ότι υπάρχει βούληση να, ξανοί... αυτό το φάκελο και επί τη βάση της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσαμε ενδεχομένω να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις για να ε, ικανοποιήσουμε τις βασικές ανησυχίες ε, όπως ε, προέκυψαν στην Ολομέλεια. Αυτό το νέο άνοιγμα αυτή η νέα βούληση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα δεδομένο και επίσης δεν είχε ε, τι, μετά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια τη δυνατότητα η Επιτροπή μας να επανεξετάσει το θέμα στο μεταξύ. Οπότε, ο στόχος σήμερα είναι να κάνουμε μια απλή ανταλλαγή απόψεων και επί τη βάση των σημερινών συζητήσεων, αφού ακούσουμε την παρουσίαση της εισηγήτρας και αφού ακούσουμε όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους, θα δούμε εξετάσουμε υπό ποιε συνθήκε θέλουμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτή την ε, έκθεση, είτε να ψηφίσουμε ε, το Σεπτέμβριο, στην επόμενη Ολομέλεια δηλαδή, είτε να ε, επιλέξουμε ένα διαφορετικό δρόμο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε ποια συνέχεια θα δοθεί. Θα αποφασίσει ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Ελπίζω να κάλυψα τι ανησυχίε του κυρίου Σέρκας και δίνω το λόγο στην κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω επίσης ε, και για τη διευκόλυνση που μου κάνετε για την ημερήσια διάταξη. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους για αυτή την αλλαγή, αλλά πιστεύω ότι όλοι μας λίγο πολύ θα χρειαστεί να πάμε ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές συνεδριάσεις. Πρόκειται για ένα θέμα ε, πολύ ενδιαφέρον, ε, παθιασμένο θα έλεγα. Στις 5 Μαΐου η Ολομέλεια απέρριψε την έκθεση. Επομένως, ε, η έκθεση αυτή απεστάλλει ξανά στην Επιτροπή ε, για την οδηγία για την οργάνωση των χρόνων εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Από τις 23 Μαρτίου του 2005 το πεδίο εφαρμογή οδηγία έχει επεκταθεί και στις οδικές μεταφορές. Και θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα που αφορά στο χρόνο εργασίας. Ε, το θέμα έχει ως εξής. Ακόμα και στο Συμβούλιο οι ενστάσεις είναι πάρα πολύ λίγες. Υπάρχουν πάρα πολύ λίγες επιφυλάξεις. Επομένως φαίνεται ότι κοντεύουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για την οδηγία. Πρόκειται για την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Ε, συνεργαστήκαμε μαζί με τον συνάδελφο Θέρκας, μαζί με, και με κάποιους άλλους συναδέλφους. Ε, παλέψαμε από κοινού στις διαπραγματεύσεις για αυτή την οδηγία με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε ότι δημιουργεί πολλές ε, αμφισημίες αυτό το, θέμα και ο κύριος Σέρκα θα θυμάται ότι εγώ συμφωνούσα να βασιστούμε στην πείρα των νέων κρατών μελών. Όντω, δεν υπάρχει πραγματική ισορροπία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη σε αυτές τις χώρες, γι' αυτό ακριβώ και χρειαζόμαστε νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και κάτι επιπλέον. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να διανοηθούμε καν ότι ο εργαζόμενος, ο, ο είναι κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του. Ε, η οδική ασφάλεια είναι και κάποιο ακόμα, ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο. Η οδηγία αυτή επεκτάθηκε και στους ιδιώτες οδηγούς ακριβώς για να διασφαλίσουμε και την οδική ασφάλεια. Στην οδηγία του 2006 γίνεται μια πλήρης ρύθμιση του ωραρίου εργασίας, του χρόνου εργασίας. Εδώ όμως αναφερόμαστε στο χρόνο εργασίας μόνο όσων ε, εκτελούν κινητές δραστηριότητες. Ε, δηλαδή δεν μιλάμε για φόρτωση, εκφόρτωση, τέτοια πράγματα. Μιλάμε για τέτοιας μορφής οδικές μεταφορές. Στην έκθεση ε, ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή να μας παρουσιάσει μια νέα πρόταση. Στο μεταξύ στο Συμβούλιο υπήρξε συμφωνία, ε, δόθηκε η συμφωνία ακόμα και από αυτούς οι οποίοι είχαν αμφισβήτηση. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι. Αν ξαναστείλουμε στην πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι να το σκεφτείτε γιατί είναι σοβαρό. Αν το ξαναστείλουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελοχεύει ο κίνδυνος η Επιτροπή να ξεκινήσει 27 διαδικασίες επί ε, Δεν υπάρχει ούτε ένα κράτος μέλος που να έχει διευρύνει το πεδίο εφαρμογής ε, αυτής της οδηγίας και ε, στις ε, οδικές μεταφορές και στους ιδιώτες. Σήμερα υπήρξε μία συνεδρίαση των συνδικάτων για να αποφασίσουν για μία κοινή θέση και από εκεί και πέρα να την αποστείλουν στο Συμβούλιο. Αν εφαρμόσουμε τον κανονισμό όσο έχει αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορέσουμε να τροποποιήσουμε την έκθεση. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε λοιπόν είναι ή να απορρίψουμε πλήρως την πρόταση ή να την εγκρίνουμε στο σύνολό της. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ακόμα, επειδή λοιπόν δεν έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε την πρόταση, θα βρεθούμε ενώπιον τη εξή κατάσταση. Όπω σα είπα και πριν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει 27 διαδικασίε παραβάση και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι προ το συμφέρον κανενό. Θα ήθελα λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, να σταθμίσετε λίγο την κατάσταση και θα ήθελα να ζητήσω και από του συντονιστέ να, δει, να δουν λίγο τη διαδικασία, να σκεφτούν ακριβώς τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε. Αν υπήρχε η δυνατότητα να τροποποιήσουμε την ίδια την οδηγία, ας πούμε, ώστε να γίνει αποδεκτή από όλους με κάποιους συμβιβασμούς, ε, με τη συνδρομή και των ε, οδηγών, των ίδιων και των συνδικάτων τους. Ε, όλα αυτά τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε μία έκθεση την οποία δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε. Προτείνω λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια έκθεση νέα καινούρια, η οποία θα μπορέσει να μας οδηγήσει σε ένα νέο συμβιβασμό, σε μια νέα συνένεση και να ξεκινήσουμε από εκεί. Θα ήθελα τώρα να σας πω το εξής. Αν δεν κάνουμε τίποτα, δηλαδή αν το πεδίο εφαρμογή οδηγίας διευρυνθεί και για τους ε, ιδιώτες, οι δαπάνες για τους ελέγχους θα ξεπεράσουν κατά πολύ τις δαπάνες που έχει προβλέψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, μεταφορά από, το, από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο, ας πούμε, σε όλες τις Ολομέλειες. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξουμε τους ιδιώτες μεταφορής. Ακριβώς και γι' αυτό λοιπόν το φαινόμενο ε, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε λίγο τη θέση μας. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Euh, σας προτείνω ε, δεδομένου του ιδιάζοντος, ας το πω έτσι, πλαισίου, εφόσον επανεξετάζετε τώρα η έκθεσή σας, σας προτείνω να ακούσουμε ευθύ αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. <clears throat> Αντίθετα με ότι ήθιστε, γιατί έτσι οι συναδελφοί μπορούν να εξακριβώσουν επί τη βάση αυτή της πρόταση που κατά τη γνώμη μας δεν λαμβάνει υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου. Να δούμε λοιπόν πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει ε, το ζήτημα. Ο Γενικός Διευθυντής, ε, ο κύριος Γκριό Πασκοαρέλη θα μας εξηγήσει τι ακριβώς μπορεί να τροποποιηθεί από την πρόταση της Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν σας εξηγήσω τι μπορεί να τροποποιηθεί στην πρόταση, θα ήθελα να υποφεληθώ από αυτή την ευκαιρία που έχω σήμερα, γιατί δεν έχω βρεθεί ε, στην Επιτροπή σας ε, τώρα τελευταία. Θέλω να σας εξηγήσω, λοιπόν, γιατί υποβαλα αυτή την πρόταση και θα μιλήσω στα αγγλικά. Η θέση της Επιτροπής και ε, αυτή η πρόταση, λοιπόν, δεν είναι ούτε αντικοινωνική ούτε ιδεολογικού χαρακτήρα. Έχει πρακτικό χαρακτήρα. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μία ε, αποτελεσματική ναι, και υλοποιήσιμη νομοθετική πράξη. Η οδηγία για το χρόνο εργασίας ε, είναι λέξη specialis ε, σε σχέση με την οδηγία, γενική οδηγία για τα ωράρια εργασίας, η οποία δεν εφαρμόζεται στους αυτοαπασχολούμενους. Αυτός ο αποκλεισμός ποτέ δεν ε, σαν φιλεγόμενο θέμα στις συζητήσεις ε, που έκαναν ε, κυρίως το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τελευταία εκδοχή της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. τώρα, για τους κινητούς εργαζόμενους ε, είναι διαφορετική κατάσταση. Γιατί όταν εγκρίθηκε η οδηγία το 2002, ε, μιλούσαμε για τους αυτοαπασχολούμενους εκτελούντους σε κινητές δραστηριότητες, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί προσωρινά. Ε, το 2009 έγινε αυτό. Και ε, η Επιτροπή έπρεπε να κάνει μια πρόταση. Είτε για τις ρυθμίσεις για την συμπεριλαβή αυτών των εργαζομένων ή για τον ολικό αποκλεισμό των μετακινούμενων εργαζομένων. Οπότε, η πρόταση που υποβάλαμε ε, συμμορφωνόταν πλήρως με τις επιλογές που εδόθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008 από τον νομοθέτη, τον Ευρωπαϊκό Νομοθέτη. Για δύο λόγους ε, κάναμε την επιλογή που κάναμε. Πρώτον, είπαμε για να είναι αποτελεσματική και υλοποιήσιμη νομική πράξη. Και ο δεύτερος λόγος είναι διότι κατά τη γνώμη μας, για την οδική ασφάλεια δεν υπήρχε κανένας βασικός λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε τους αυτοαπασχολούμενους ε, στην οδηγία. Ας θα σχολιάσω το δεύτερο, το δεύτερο αυτό λόγο πρώτα. Όπως είπε και η συγγύτρια κυρία Μπάουερ, από το 2002 και μετά έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες για τον χρόνο οδήγησης και για τον χρόνο ανάπαυσης εφαρμόζονται σε όλους οι κανόνες, για του, εφαρμόζονται και για τους αυτοαπασχολούμενους και για τους μισθωτούς και δεν είναι μόνο αυστηρή, αλλά εφαρμόζονται και αυστηρά, γιατί μέσα σε όλα τα φορτηγά πρέπει να υπάρχει ε, ψηφιακός ταχυγράφος, ε, δηλαδή είναι ένα μηχάνημα ε, το οποίο είναι υδατοστεγές εισαγωγικά μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου που είναι υποχρεωτικό ε, για όλα τα φορτηγά και υποχρεώνουν τους οδηγούς να έχουν χρόνο ανάπαυσης ε, συγκεκριμένα. Δηλαδή συνεχίζει να ε, γράφει, να καταγράφει τα δεδομένα η μηχανή και γίνονται περιοδικοί έλεγχοι. Τώρα, 80 με 90% του χρόνου εργασίας των μετακινόμενων εργαζομένων είναι η οδήγηση. Το ίδιο και για τους αυτοπασχολούμενους και για τους μισθωτούς. Οπότε με αυτό τον κανονισμό το 2006 καλύψαμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον χρόνο εργασία και όχι μόνο τον χρόνο οδήγηση, αλλά και το χρόνο εργασία όλων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων. Το επιχείρημα αυτό περιοδικής ασφάλειας δεν βασίζεται, δεν ε, επαληθεύεται από τις στατιστικές και από τις μελέτες που κάναμε πριν υποβάλουμε την πρότασή μας. Έχουμε μια στατιστική βάση δεδομένων για την οθική ασφάλεια. Χρησιμοποιήσαμε και μια μελέτη που έγινε από έναν ανεξάρτητο σύμβουλο, που λέγεται η εταιρεία, και όλα τα στοιχεία, όλες οι μελέτες δείχνουν, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα φόρτιγα εμπλέκονται μόνο σε 6% του συνόλου των ατυχημάτων. Εμπλέκονται, δεν ευθύνονται για το 6% των ατυχημάτων. Και η κόποση είναι ε, βασική αιτία μόνο στο 6% αυτού του 6% των ατυχημάτων. Δηλαδή 0,4% και λιγότερο του συνόλου των ατυχημάτων μπορούμε να αποδώσουμε ε, στην κόποση ως βασικό λόγο. Οπότε η ρύθμιση του χρόνου εργασίας ε, επί τη βάση αυτής ε, λόγου να κατοχυρώσουμε την οδική ασφάλεια ε, είναι κάτι το υπερβολικό σε σχέση με τις ανάγκες μας. Δείχνει η μελέτη ότι η κόποση δεν σχετίζεται μόνο με τις ώρες εργασίας. Ε, το πιο επικίνδυνο είναι η χρόνια κόπωση που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, ε, όπως παραδείγματο χάρη προβλήματα υπνίας, άλλα προβλήματα υγεία, ε, υγείας, αλκοόλ, κάπνισμα, ναρκωτικά ε, και κάποιες κάποιοι τρόποι ζωής ε, που ε, είναι επιβλαβή το ίδιο και για του αυτοαπασχολούμενου και για τους μισθωτούς. Τώρα να, να προσθέσουμε άλλη μια νομική πράξη για το χρόνο εργασίας ε, για τους μετακινούμενους εργαζόμενου για να ενισχύσουμε την οδική ασφάλεια. Δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν έχουμε στοιχεία να στηρίξουμε μια τέτοια κίνηση. Και τώρα επανέρχομαι στη, στην πρώτη αιτία υποβολή πρόταση, στην υλοποιησιμότητα τη νομική πράξη. Ε, στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολο, για να μην πω αδύνατο, να ελέγξουμε το χρόνο εργασίας των αυτοαποσχολουμένων. Δεν μπορούμε να βάλουμε ψηφιακό ταχυγράφο στα γραφεία τους ή στα σπίτια τους για να ελέγξουμε για πόση ώρα εργάζονται. για να είμαστε σοβαροί όταν νομοθετούμε, δεν μπορούμε να εκπονούμε νομικέ πράξει που δεν είναι υλοποιήσιμε. Πρέπει ε, μάλλον να εφαρμόσουμε αυτά που υπάρχουν ήδη για το χρόνο οδήγησης και για το χρόνο ανάπαυσης για τις σχετικές οδηγίες. Εργάζεται εντατικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή αυτών των δύο νομικών πράξεων και είπαμε ισχύει και για τους αυτοπασχολούμενου και για τους μισθωτούς και πρέπει να απλουστεύσουμε την νομοθεσία, να μην έχουμε υπερβολικό διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις. Πρέπει να ενισχύσουμε και τους ελέγχους για όσους υπάγονται στην οδηγία χρονοεργασίας, κυρίως για τους ψευδοαπασχολούμενους, όπως ονομάζονται και που τους περιέγραψε η κυρία Μπάουερ, η συγγετριά μας. Το τωρινό κείμενο αφήνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν η οικία νομοθεσία στους αυτοαπασχολούμενους. Δεν αποκλείεται αυτό στο κανονισμό. Τώρα ας δούμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν για την επανεξέταση του ζητήματος. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που μας είπε η κυρία Μπαουρά, αν κατάλαβα καλά τι είπε, γιατί δεν μιλώ ογκρικά. Είπε λοιπόν ότι προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα, να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση. Το ETF, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Οδικών Μεταφορέων, συνεδριάζει σήμερα και αύριο, ξέρετε, για αυτή την απόφαση. Και περιμένουμε να δούμε τι έχουν να πούν οι κοινωνικοί εταίροι. Μας ενδιαφέρει και σίγουρα και η δική σας η Επιτροπή το ίδιο θέλει. Ε, ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οδικών Μεταφορέων ε, να δούμε μετά αφού έχουμε αυτά τα στοιχεία ποιες δυνατότητες επανεξέτασης υπάρχουν εμείς προτιθέμεθα να συνεργαστούμε επικοδομητικά με το Κοινοβούλιο, με το Συμβούλιο, με τους κοινωνικούς εταίρους για να βρούμε μια λύση. Το σημαντικό για μας είναι πρώτον να μεριμνήσουμε ώστε ο νομοθέτης θα εκπονήσει ε, εφαρμόσιμες νομικές πράξεις και δεύτερον θα εκπονήσει νομοθεσία που δεν αιτιολογείται ή μάλλον που βασίζεται σε πραγματικές αιτίες. Δηλαδή, ε, άμα επικαλεστούμε την οδική ασφάλεια, αυτός να είναι ο ουσιαστικός λόγος, όχι να χρησιμοποιηθεί ε, ως ε, ψευδής ε, λόγος και επίσης να αποφύγουμε και το υπερβάλλον διοικητικό άχθος. Μάλιστα ε, κύριε Γενική Διευθυντά, αλλά δεν απαντήσατε στην ερώτηση μου φαίνεται. Δεν μας είπατε τι θα αιτιολογούσε το να ξανανοίξουμε το φάκελο. Περιγράψτε μια κατάσταση που δείχνει ότι θα μπορούσαμε και να δεν το ξανανοίξουμε το φάκελο, αλλά δεν μας δώσατε συγκεκριμένε αιτίε. Αναφερθήκατε στατιστικά στοιχεία για την ασφάλεια, που μας δίνουν την εντύπωση ότι οι οδηγοί των φορτηγών, των βαρέων οχημάτων, ε, δεν έχουν μια συμπεριφορά επικίνδυνη όταν οδηγούν, ε, δεν ευθύνονται για τα, σε μεγάλο βαθμό για τα ατυχήματα, αλλά ε, έχουμε και τους μισθωτούς. Και είπατε ότι καλύπτουμε και τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους. Μα η ουσία του κειμένου είναι η διάκριση ανάμεσα στους, στις δύο κατηγορίες. Δηλαδή θα έχουμε αυστηρότερους κανόνες για τους μεν σε σχέση με τους δε. Σας ξαναδίνω το λόγο σας παρακαλώ για να μας πείτε συγκεκριμένα ε, ε, περί πρόκειται, γιατί η τάση μας ήταν να επιβεβαιώσουμε αυτή τη ψηφοφορία, γιατί ο Επίτροπος ήθελε να μας πει ότι μετά τις διαβουλεύσεις με διάφορους εταίρους ε, θα πρέπει να επανεξετάσουμε κάποιες πτυχές του ζητήματος. Μα ποιες είναι οι πτυχές του ζητήματος, εφόσον τα στατιστικά στοιχεία, ξέρετε, τα ερμηνεύουν και τα κάνουμε να λένε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι λόγος αυτός. Μπορείτε να μας πείτε, επί τη βάση της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επί ποιας βάσεως θα μπορούσατε να λάβετε υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου που δεν μπορεί να δεχτείτε τον αποκλεισμό από το πεδίο εφαρμογής οδηγίας των αυτοαποσχολουμένων. Madame, euh, les... Οι οδηγοί είναι άνθρωποι όπως και όλοι οι άλλοι, επαγγελματίες. Διακόπτη πρόεδρος, με συγχωρείτε, ε. με συγχωρείτε. Ε, πείτε μου πολύ συγκεκριμένα για ποιο λόγο πρέπει να ξανανοίξουμε το θέμα αυτό. Ε, madame, ε, la commission... Κυρία μου, η Κομισιόν έχει κάνει την πρότασή της. Το Κοινοβούλιο πρέπει να επιβεβαιώσει ή όχι τη ψηφοφορία που έγινε στην περασμένη θητεία. Σας είπα ότι οι κοινωνικοί εταίροι συζητούν το θέμα αυτό. Άκουσα, αν κατάλαβα καλά, την κυρία Μπάουερ να λέει ότι ε, μπορεί να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση. Εγώ λέω ναι βεβαίω να γίνει, να την ακούσουμε για να... και θέλουμε να ακούσουμε και του, τι θα πούνε οι κοινωνικοί εταίροι αύριο. Επαναλαμβάνω, η θέση της Κομισιόν είναι είμαστε ανοιχτοί και σε άλλες λύσεις. Δεν τις γνωρίζω ακόμη, αλλά οποιαδήποτε λύση άλλη θέλετε να συζητήσουμε θα πρέπει να ε, μας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε σαφώς την νομοθεσία αυτή χωρίς να δημιουργείται ε, ε, να δημιουργείται επιπλέον νομοθετικός και διοικητικός φόρτος εκεί που δεν υπάρχει ανάγκη. Πρόεδρος, ο κύριος Ροζέ ζήτησε το λόγο ή μάλλον θα δώσω το λόγο πρώτα πρώτα στον κύριο Σερκάς που α, αντικαθιστά τον κύριο Σερκιούς. Madame Brarkin, donc vous aurez la parole ensuite. Euh, κυρία Μπρανκίν θα πάρει μετά το λόγο. Αρχίζουμε τον κύριο Σερκάς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε θα μιλήσω εξ ονόματος του Στίβεν Χιούζ, ο οποίος ήταν εισηγητής της ομάδας μου για το θέμα αυτό και θα μιλήσω και εξ ονόματος της ε, ομάδας των σοσιαλιστών. Θα ξεκινήσαμε τη συζήτηση αυτή με μια επιβεβαίωση δική σας κυρία Πρόεδρε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φαντάζομαι και ο Επίτροπος Σπίτλα είχε επιδείξει την καλή διάθεση να βρούμε ένα συμβιβασμό και να βρούμε και μια άγουσα για το συμβιβασμό. Αλλά μόλις ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι ο Επίτροπος Σπίτλα βέβαια, ε, αλλά δεν είναι αυτά που μας υποσχέθηκε. Ε, το παίζουμε πολύ καιρό αυτό το ε, παιχνιδάκι είναι απασχόληση. Είναι ο Επίτροπος Ταγιάννη ο υπεύθυνο, όχι ο κύριος Σίτλα. Τέλος πάντων, ακόμα περισσότερο με διευκολύνεται, κυρία Πρόεδρε, διότι συνέχεια μας κάνουν δηλώσεις τις οποίες ε, στην πράξη δεν υλοποιούν. Προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρόνο, μα τάζουν ότι θα ξανανοίξει το θέμα και θα κάνουμε νέε διαπραγματεύσει και αυτό δεν γίνεται ποτέ. Όσον αφορά τώρα για τη συζήτηση με του κοινωνικού εταίρου, ε, μας λείπουν λίγε ώρες για τη, για συνάντηση. Εγώ μίλησα με του κοινωνικούς εταίρους και μας λένε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βασική θέση που είναι η συμπερίληψη των αυτοαπασχολουμένων. Ακούσαμε κυρία Πρόεδρε, κατά την άποψή μου είναι μάλλον σκάνδαλο αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να φρονεί ότι η κούραση δεν έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια προσπαθούμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο το 2002 έτυχε συνένεση από την αντίθετη ένωση. Η οδηγία το 2002, αντίθετα με αυτό που μας είπε ε, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, ε, είχε δύο χώρες οι οποίες ήταν κατά, τη Φιλανδία και την Ισπανία, τη χώρα μου, και όλοι αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε τους αυτοαπασχολούμενους για λόγους υγείας και ασφάλειας για τους οδηγούς μας και για τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι οδηγούν στους δρόμους. Σήμερα διαπιστώνω εδώ με έκπληξη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται ότι υπάρχει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ κούρασης και ε, των ε, τροχαίων ατυχημάτων και η οδηγία για το χρόνο εργασία δεν συμπεριλαμβάνει σε αυτό αποσχολουμένου και αυτό μα το χρησιμοποιείται σε επιχείρημα. Δεν μα περιλαμβάνονται διότι είναι διαφορετικό ε, για αυτού που δεν οδηγούν και αυτού που οδηγούν ε, το θέμα. Και επίση αυτό που είναι σκάνδαλο είναι ότι μα επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να διαχειριστούμε και να ξέρουμε τι κάνουν οι αυτοαποσχολούμενοι στο σπίτι του ή στο γραφείο του, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο χρόνο εργασία ο οποίο λαμβάνουμε υπόψη δεν είναι αυτό ε, του γραφείου ή του σπιτιού, ο οποίο είναι εκτό πεδίου εφαρμογή οδηγία. Ο οποιο λαμβανουμε υποψη δεν ειναι αυτο του γραφειου η του σπιτιου ο οποιο ειναι εκτο παιδι εφαρμογη οδηγια ο χρονο που προσμετράται για να δούμε την κούραση είναι η φυσική προσπάθεια όταν οδηγούν ή όταν μεταφέρουν κάτι. Όχι όταν διαχειρίζονται το γραφείο του ή ό,τι κάνουν στο σπίτι του. Ζητώ συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, δεν θα καθυστερήσω άλλο αλλά δεν νομίζω ότι είναι κανείς διατεθειμένος να κάνει επικοδομητικό διάλογο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έσπασε τη συνένεση που υπήρχε μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έσπασε αυτή τη συνένεση και διακυβεύεται αυτή τη στιγμή η υγεία και η ασφάλεια των αυτοαπασχολημένων οδηγών αλλά και των πολιτών που κυκλοφορούν στους δρόμους γιατί μπορεί να υπάρχουν οδηγοί που θα είναι εξαιρετικά κουρασμένοι. Και πάντα χρησιμοποιούν το άλοθη και μας λένε ότι αυτό είναι ένας κανονισμός ο οποίος ε, θα οδηγήσει σε μεγάλη γραφειοκρατία. Όταν στην πράξη το να συμπεριλάβουμε τους αυτοαποσχολημένους ουσιαστικά θα, θα πάρα πολύ τη γραφειοκρατία. Οι ψευδοαποσχολούμενοι και αυτοαποσχολούμενοι ε, είναι μια γραφειοκρατική κατάσταση η οποία θα είναι χωρίς τέλος, αλλά εάν υπόκεινται όλοι στις ίδιες διαδικασίες, ε, στις ίδιες, στους ίδιους κανονισμούς, θα διευκολυνθεί η δουλειά μας. Διότι... Ε, δεν θα χρειάζεται ένας ε, ε, συνοριοφύλακας, για παράδειγμα, στην Ισπανία, όταν συναντά ένα Πολωνό να ξέρει αν είναι αυτοαπασχολούμενος ή ψευδοαπασχολούμενος. Ούτε θα τον ενδιαφέρει αν εργάζεται για κάποια επιχείρηση ή αν είναι αυτοαπασχολούμενος. Δεν χρειάζεται καν οδηγία για το χρόνο εργασίας. Υπάρχουν οδηγίες για το χρόνο εργασίας, υπάρχουν και για κάθε μία από τις τάσεις και τις δράσεις που ε, αφορούν στην νομοθεσία και τις παραβάσεις. Το να εφαρμόσουμε ένα κανόνα ε, ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να ξέρουμε τις βασικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Δρόμη, ό,τι και να λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι, στο, ε, είναι έρμεο της κούρασης των οδηγών. Και αν δεν ρυθμίσουμε αυτή την κατάσταση, δεν θα λυθεί το θέμα. Αύριο θα την ψηφίσουμε αυτή την απόφαση. Το Κοινοβούλιο τρεις φορές είπε ότι αυτή η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να απορριφθεί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο για να μην κάνουν αυτό που πρέπει. Θα τους πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όλους όσους δεν τηρούν τον νόμο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Άρκιν, την επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση, λένε και κάποιοι ότι χάνουμε το χρόνο μας εδώ, δεν ξέρω. Εγώ όμως συμφωνώ να μην έχουμε υπερβολική νομοθεσία για κάποιους ε, εργαζόμενους. Ε, εγώ νομίζω ότι δεν είναι χάσιμο χρόνο. Εν πάση περιπτώσει να σας δώσω τη δική μου τη θέση και τη θέση ξέρετε τη θέση της ομάδας μου του περασμένου Απριλίου, η οποία ήταν ομόφωνη. Εδώ μιλάμε για χρόνο εργασίας. Και βεβαίως υπάρχει η 561 του 2006 και υπάρχει και ο ψηφιακό ταχυγράφο, όπω είπε και ο κύριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ξέρουμε ότι 80 με 90% του χρόνου εργασία, ακόμη και των αυτοαπασχολούμενων, είναι χρόνο οδήγηση. Άρα λοιπόν κάτι κάνει αυτή η οδηγία του 2006, παρόλο που δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση. Ε, αν δούμε λιγάκι τα θέματα οδικής ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε κάποια συγκεκριμένη δημοσκόπηση που έγινε ε, μας είπε ότι τα φορτηγά ε, ήταν ε, μπλέκονταν στο 6% μονάχα των ο, τροχαίων στοιχημάτων αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι το ποσοστό μεταξύ του συνόλου των οχημάτων που μελετήθηκαν που προσωπούσαν τα φορτηγά. Μπάση περιπτώσει υπάρχουν και άλλες ε, μελέτες που ένα παραδείγματο χάρη, μια παραδείγματο χάρη από τη Φινλανδία που λέει ότι το 25 25% των ατυχημάτων οφείλονταν στους οδη, που έγιναν οφείλονταν στους οδηγούς των φορτηγών. Αυτό είναι το αντίθετο από αυτό που ακούσαμε τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Άρα τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Τώρα ε, η Κομισιόν α, ε, είπε ο κάποιος προηγούμενος συνάδελφός μας ότι θεωρεί ότι η Κομισιόν ε, ότι η κόπωση δεν είναι η αιτία των δυστυχημάτων. Συγγνώμη, βεβαίως η Κομισιόν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό τη. Εγώ απλώ αναρωτιέμαι έστω ότι κάνουμε μια νομοθετική πράξη για την κόπωση. Θα βελτιώσουμε τα πράγματα. Είναι, θα είναι αδύνατο να εφαρμοστεί ε, μια τέτοια νομοθετική πράξη. Θα γελιοποιηθούμε και όλα και πολύ αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί και πολλοί επιχειρηματίες θα θεωρήσουν άχρηστο αυτό το, άχρηστη αυτή την νομοθετική πράξη. Αν είχαμε σίγουρα επιδεικτικά στοιχεία που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μπορεί να κάναμε κάτι. Αλλά ε, τώρα επειδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κάτι την οποία τα πράγματα είναι ακόμη φλού και δεν υπάρχει σαφής γραμμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Πρόεδρο κτλ. Εγώ θα έλεγα να συμφωνήσουμε με την εισηγήτρια και να ξεκινήσουμε τη δουλειά για μια καινούρια έκθεση. Η κυρία Εμιλή Τουρίνεν. Ναι, Είμαι Φινλανδέζα και θα μιλήσω Φινλανδικά. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν σοβαρότατες ε, διαφορές απόψεων. Έχουμε τελείως διαφορετική φιλοσοφία σχετικά με το τι σημαίνει οδική ασφάλεια, έχω την εντύπωση. Ε, το Μάιο Έγινε ψηφοφορία στην ε, ε, Ολομέλεια και πιστεύουμε ότι αυτή η ψηφοφορία δεν μπορεί να γνωριθεί. Δόθηκαν σαφή μηνύματα σε εκείνη την ε, ψηφοφορία και εκπλησόμεθα που επανέρχεται εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αμφισβητεί την ε, ψηφοφορία αυτή. Μας λέει επίσης η Κομισιόν ότι συζητούν αυτή τη στιγμή ε, οι κοινωνικοί εταίροι. Εγώ νομίζω ότι δεν γίνεται συζήτηση μεταξύ κοινωνικών ε, εταίρων ε, και οι αυτοαπασχολούμενοι δεν θα πρέπει να αποκλειστούν. Πρόεδρος, υπάρχουν άλλοι 11, 12 ε, ομιλητές. Monsieur Roger Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι σε μια περίεργη και ασυνήθιστη κατάσταση. Συμφωνώ με τη θέση του εργατικού κόμματο τη κυβέρνηση ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτι που μου συμβαίνει πάρα πάρα πολύ σπάνια. Προηγούμενα είπα ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλέ νομοθετικέ πράξει και αυτό δεν το θέλουμε. Ε, Ακριβώ. Να ένα παράδειγμα εδώ. Δεν θέλουμε να υπάρξουν επιπλέον κανόνε. Δεν θέλουμε να υπάρξουν και άλλα επίπεδα νομοθεσία πέρα από τα εφιστάμενα. Η θέση τη Βρετανική κυβέρνηση κυβέρνηση είναι ότι πρώτον θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί η οδηγία του χρόνου εργασίας στους αυτοαπασχολούμενους και δεύτερον ότι υπάρχουν αρκετές νομοθετικές πράξεις που ρυθμίζουν τα προβλήματα αυτά ξέρω, ίσως ο κύριος Σέρκας να θέλει, να, πρέπει να έρθει, να παρακολουθήσει, να ζήσει μια-δυο εβδομάδες ε, το, ένα φορτηγατζί στη, ανά την Ευρώπη για να σημειώνει τι γίνεται. Δεν ξέρω και αντιστοίχω να ε, πάμε να παρακολουθήσουμε και τον κύριο Σέρκας ε, τι κάνει στη δουλειά του και πόσες ώρες οδηγεί ο ίδιος. Πολλέ ώρες φαντάζομαι και εγώ και εγώ οδηγώ πάρα πολύ τέλος πάντων το κόμμα μου είναι κατά της ε, του χρόνου εργασία, γι' αυτό θέλουμε να αποχωρήσουμε και από την Ευρώπη τελικά επουδενή λόγο πάντως θέλουμε επέκταση τη της του χρόνου εργασίας και κυρία Πρόεδρε σα παρακαλώ ας αφήσουμε κατά μέρο την ασφάλεια η ασφάλεια, η οδική ασφάλεια είναι ε, είναι δευτερεύον παράγοντας. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο κάναμε μία μελέτη και είδαμε ότι 50% των αλλοδαπών φορτηγών έχουν προβλήματα τεχνικά. Λοιπόν, ας αφήσουμε την οδική ε, ασφάλεια και τους ελέγχους ε, στους φορτηγατζίδες και ας κοιτάξουμε να δούμε από τεχνικής απόψεως και από μηχανικής απόψεως πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ξέρετε, μία πρόεδρος επιτροπής ε, δεν έχει και τόσες πολλές εξουσίες ε, και δεν μπορώ να ε, ευθύνομαι εγώ για αυτά που λένε τα μέλη της επιτροπής. Κυρίως θα μιλάμε για την ασφάλεια. Ευλήν Χαγκνέρ και ο κύριος Τόμας Χάντελ ακολουθούν. Η κυρία Ρέγνερ πρώτη. Το κατά πόσον ένας φορτηγατζής που ταξιδεύει στην Ευρώπη είναι αυτοαπασχολούμενος ή όχι ή κατά πόσον είναι μισθωτός. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαπιστώσουμε. Ε, τουλάχιστον για την Αυστρία αυτό ισχύει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρούμε. Άρα λοιπόν όλοι οι μισθωτοί αυτοαπασχολούμενοι ή όχι θα πρέπει να την χάνουν της ίδιας μεταχείρισης. Αυτό σαν πρώτη σκέψη. Τώρα για την οδική ασφάλεια βεβαίως ξέρω ότι αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα αλλά ε, ε, κάθε χρόνο έχουμε 100 θύμα, 100 ζωές που χάνονται στο το χρόνο στην Αυστρία επειδή κοιμάται για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου άνθρωπος αυτός. Μεταξύ αυτών των 100 θυμάτων είναι και πάρα πολλοί οδηγοί φορτηγών. Λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς που λένε ότι η κόποση δεν ε, οδηγεί σε ατυχήματα ή δυστυχήματα. Και δύο λόγια ακόμη για την επιπλέον γραφειοκρατία ή επιπλέον επίπεδο νομοθετικών πράξεων κτλ. Και ε, δεν θέλουμε να διχάσουμε τους οδηγούς φορτηγών. Ε, άρα καλύτερο είναι ούτε επιπλέον γραφειοκρατία να κάνουμε ούτε κάτι το ιδιαίτερο για τους αυτοαποσχολούμενους. Λοιπόν, ο, ίση μεταχείριση για όλους και η ίδια νομοθετική πράξη για όλους. κύριος Τόμας Χάντελ και κυρία Λίζα Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τόμας Χέντελ λέγομαι, όχι Χάντελ. Υπάρχουν και δύο βουλίτσες πάνω από το Α στο όνομά μου. Λοιπόν, είμαι Γερμανός συνδικαλιστής και θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την Επιτροπή αυτή ε, και το Κοινοβούλιο γενικότερα για τη δουλειά που έκανε στην περασμένη θητεία ε, για το έργο το οποίο έκανε για την, σχετικά με το χρόνο εργασίας όπου δεν επιδεινώθηκαν τα πράγματα όπως θα μπορούσαν να είχαν επιδεινωθεί αν δεν δουλεύατε εσείς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα. Τώρα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι κατά της οποιασδήποτε τροπολογίες της μέχρι του οδηγίας. Δεν υπάρχει λύση, όλη η συμμεταχείριση δεν αλλάζουμε τίποτα. Τώρα και κάτι τι άλλο να πω. Ήμουν δικαστής σε ένα εργατικό δικαστήριο στη χώρα μου πριν από μερικά χρόνια και ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο χρόνο, πόση δουλειά χρειάζεται για να διαπιστώσουμε αν κάποιος είναι αυτοαπασχολούμενος ή όχι ή όχι. όπω προτείνει η Κομισιόν να κάνουμε κάτι ε, ιδιαίτερο ε, ε, και το ότι υποθέτει η Κομισιόν ότι είναι αρκετά απλό να χωρίσουμε τους μεν από τους δε είναι για μένα ουτοπία. Ε, ε, η, δεν είναι λόγο μπορώ να συμφωνήσω με την θέση αυτή. Και θα ήθελα να κάνω και μια τρίτη παρατήρηση σχετικά με αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν που μίλησε για τις επιχειρήσεις, για τους επιχειρηματίες. Κοιτάξτε, θα, εγώ θα αντιστρέψω το επιχείρημα που είπε η Κομισιόν. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να μην παραφορτώσουμε τους εργαζόμενους. Το, όταν κάποιος έχει δουλέψει πολλά χρόνια, να τον βάλουμε να δουλεύει και πάρα πολλές ώρες, είναι υπερβολικό. Νομίζω ότι για να μπορέσει κανείς να ανταποκριθεί σε τεράστιο ωράριο εργασίας, ιδιαίτερα μετά από πολλά χρόνια δουλειάς, θα πρέπει να προσφύγει σε άλλου είδους μέσα και ναρκωτικά ενδεχομένως. Λοιπόν, δεν θέλουμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν θέλουμε να ε, θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία των ενδιαφερομένων εδώ και σε τελευταία ανάλυση ούτε και για τον ανταγωνισμό θα ήταν καλό να κάνουμε κάτι τέτοιο αν βγάλουμε από εδώ ορισμένους εργαζόμενους ορισμένους οδηγούς ε, θα καταλήγαμε να ε, πιέσουμε αν θέλετε να οδηγήσουμε τους υπαλλήλους οδηγούς να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι ούτως ώστε να μην ε, υπόκεινται στην οδηγία αυτή και να μπορούν να δουλεύουν μετά κάτω από χειρότερες συνθήκες δουλειάς. Ε, από πλευρά μου είμαι κάθετα αντίθετος με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακόμη 12 έχω λέει πρόεδρος. Κλείνω τον κατάλογο των ομιλητών και ε, θα πρέπει να μειώσω και το χρόνο αγόρευσης στα δύο λεφτά ανά άτομο. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία για κονσάρι που θα είναι η μόνη που θα πρέπει να τηρήσει τα δύο λεπτά. Τέλος πάντων δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Υπάρχει μια παρεξήγηση στον αέρα για το θέμα αυτό. Καλό θα ήταν λοιπόν να μην ψηφίσουμε και να το δούμε με την ησυχία μας λίγο το θέμα. Ο προλαλή σα μίλησε για ανταγωνισμό. Υποθέτω ότι όλοι μας στην προεκλογική μας εκστρατεία ήμασταν υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα ήταν λοιπόν τόσο κακό να υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι σας το λέω τώρα ενθερμό, αλλά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη, να τα δούμε και από αυτή την πτυχή. Να σας πω λίγο πώς έχουν τα πράγματα στη Φιλανδία. Στη Φιλανδία το 70% των ε, μεταφορικών επιχειρήσεων είναι επιχειρήσεις που έχουν ένα ή δύο φορτηγά οχήματα. Έχουμε κανονισμό για το χρόνο εργασίας και το χρόνο ε, ξεκούρασης και αν δημιουργήσουμε περαιτέρω νομοθεσία για το θέμα αυτό, θα δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Οι εκτιμήσεις μας λοιπόν στη Φιλανδία είναι ότι παρά το γεγονός ότι το κόστος είναι ήδη υψηλότερο από το μέσο όρο στην Ευρώπη, θα ξεπεράσουν, ε, θα φτάσουν σε δυσθεώρητα ύψη, ε, ειδικά σε περιοχές οι οποίες είναι αεροκατοικημένε. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξή. Υπάρχει δυνατότητα να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό, σε ένα συμβιβασμό ο οποίο θα ικανοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερου. Η συγγήτρια έχει σκεφτεί Ποιο θα μπορούσε να ήταν ε, αυτός ο συμβιβασμό, Τι άποψη έχει η συγγήτρια για ένα πιθανό συμβιβασμό. Κατανοώ και τις ανησυχίες των υπολείπων, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι βασική ανησυχία. Εμένα μου φαίνεται περίεργο εμείς ως νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να ξανακοιτάξουμε οποιοδήποτε θέμα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει ένας νέος συμβιβασμός. Και ποιος θα ήταν αυτός. Χαίρομαι που ε, έχουμε περισσότερο χρόνο. Ε, η κυρία, η κυρία Λίν και μετά η κυρία Ρουντζελή. Ευχαριστώ. Για όσου από εσά ήσασταν εδώ στην προηγούμενη θητεία, ξέρετε ότι εγώ ήμουν πάντα αντίθετη στην οδηγία για το χρόνο εργασία και πίστευα ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να επιλέγουν ελεύθερα πόσε ώρε εργάζονται. Βέβαια, πάντα έλεγα ότι αν κάποιος έχει ε, στα χέρια του και τη ζωή κάποιου άλλου, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Για τους μετακινούμενους εργαζόμενους, ε, οδηγούς φορτηγών, οδηγούς ε, μεγάλων βαρέων οχημάτων, αλλάζουν τα πράγματα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορά αν μιλάμε για αυτό απασχολούμενο ή για απασχολούμενο σε μια επιχείρημα. Αν κάποιος προκαλέσει ένα οδικό ατύχημα, μπορεί να σκοτωθούν, να έχουμε θύματα στο δρόμο και είπατε ότι ο οδηγός για το χρόνο εργασίας αυτό. Αλλά αν έχει δουλέψει μια-δυο ώρε πριν ξεκινήσει να οδηγεί, τότε θα είσαι ήδη κουρασμένο και στο τέλο τη βάρδιά σου, κατά πάσα πιθανότητα, ε, η κρίση σου δεν θα είναι και τόσο διαυγή όσο σε άλλη περίπτωση. Και χρησιμοποιήστε και το επιχείρημα ότι και οι προβουλευτέ οδηγούν. Εγώ προσωπικά γυρίζοντα από την Ολομέλεια στο Στρασβούργο δεν οδηγώ. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη για να οδηγήσω και δυόμιση ώρε μετά το αεροδρόμιο. Ε, δεν το κάνουμε αυτό. Επομένω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που χρησιμοποιούν του δρόμου και υπάρχουν και άλλοι οδηγοί. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι γίνονται αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί ακριβώ για να παρακάμψουν την οδηγία. Και λέτε και εσείς ότι θα πρέπει να διαγράψουμε ουσιαστικά την οδηγία για όλους τους ε, μεταφερόμενους οδηγούς, διότι λέτε ότι αυτοί οι οποίοι ε, εργάζονται σε επιχειρήσεις και προκαλούν αντίχημα εκεί θα πρέπει να υπάρχει νομοθεσία και για τους αυτοαπασχολούμενους δεν θα πρέπει να έχουμε καμία νομοθεσία. Δεν το καταλαβαίνω το επιχείρημά σας. Θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί όταν κάνουμε νομοθεσία. Ή θα ισχύει για όλους ή δεν θα ισχύει για κανένα. Κυρίως όταν έχετε να κάνετε και με ζωή άλλων ανθρώπων. Ε, υπάρχουν ε, οδηγοί οποίοι εργάζονται διαμεθοριακά, γι' αυτό ακριβώ και δεν θα πρέπει να κάνουμε ρύθμιση σε επίπεδο κράτου μέλου, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Λίζα Ροντζόλη και μετά ο κύριο Ματιέ Χώστ. Ζητώ συγγνώμη, πρέπει να. Μάλλον έχω σκοτώσει όλα σα τα ονόματα, αλλά είναι πολύ δύσκολα. Ναι, σα ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνδιαλεγόμεθα με, τις, ε, με τους κοινωνικούς εταίρους και όλους τους ενδιαφερομένους. Και αυτό για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση και να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε ένα συμβιβασμό. Θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει να ανοίγουμε πάντα την πόρτα στο διάλογο και να μην κλείνουμε πόρτες, ε, διότι αυτά, δεν οδηγούν, αυτά τα μέτρα δεν οδηγούν πουθενά. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη δυνατότητα που μα είπε η συγκήτρια Μπάουερ να ετοιμάσει ίσως μια νέα πρόταση και να της δώσουμε περαιτέρω χρόνο για να συζητήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ. Ματιέ και στη συνέχεια κυρία Έλληνα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Επιτροπή Μεταφορών είχα την ευκαιρία να εργαστώ για το χρόνο οδήγηση και ανάπαυση. Και ξέρετε και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέδωσαν ιδιαίτερο βάρο στο θέμα τη ασφάλεια. Και άμα δείτε για τι ώρε, γιατί εδώ μιλάμε για το ανώτατο όριο των 9 ώρων οδήγηση, 56 την εβδομάδα και 90 κατά ανώτατο όριο στι 2 εβδομάδε, δηλαδή 45 και 45. Ε, η, ο χρόνο οδήγηση και ανάπαυση είναι πολύ πιο αυστηρό από το χρόνο εργασία. Οπότε τώρα μα μιλάει για την ασφάλεια η Επιτροπή, αυτό αναφέρεται. Τα κράτη-μέλη σήμερα δεν καταφέρνουν ούτε το 2% να ελέγξουν ε, για τον χρόνο οδήγηση και ανάπαυση και σήμερα ξέρουμε ότι είναι αδύνατον να ελεγχθεί ο χρόνο εργασία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε εδώ για αξιοπιστία και όχι για ασφάλεια. Αυτό είναι το θέμα μα. Επίση ήρθα σε επαφέ ε, στην προηγούμενη θητεία και στην τωρινή θητεία με τα συνδικάτα και συμφωνούν ότι δεν γίνεται η έλεγχη και άρα πρέπει να βρούμε μία λύση. Πρέπει να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Κάτι άλλο τώρα. Μιλάμε εδώ για έναν οδηγό με 3,5 τόνους φορτηγό. Αν εγώ ε, ε, έχω 3,4 τόνους, ε, αν ζυγείς 3,4 τόνους στο φορτηγό μου, δεν υπάγομαι στους ίδιους κανόνες για την οδηγία, για την, για την οδήγηση και για την ανάπαυση. Πρέπει να δούμε αυτό το όριο των 3,5 τόνων, γιατί στην προηγούμενη θητεία εν μέρει αυτό είχαμε προτείνει, γιατί έτσι θα σημειωνόταν η κοινωνική πρόοδος και αν μιλ θέλετε ουσιαστικά να μιλήσουμε για την ασφάλεια, πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το όριο των 3,5 τόνων και τον ταχυγράφο, γιατί μόνο έτσι είναι δυνατός ο έλεγχο σε όλα τα κράτη-μέλη. Μάλιστα, σα ευχαριστούμε. Η κυρία Φιγκυρέιντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη το 2002 όταν συζητήθηκε η οδηγία που τώρα είναι σε ισχύ έγινε μια παρεμφερή συζήτηση εδώ. Ήδη από τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρηματολογούσε με τον ίδιο τρόπο. Και ε, εγώ η ίδια, και όχι μόνο εγώ και άλλοι, υπερεμήνθηκαν σε εξή θέσεως Ότι πρέπει να ρυθμίσουμε την κατάσταση για όλους και για τους αυτοαπασχολούμενους, για να αποφύγουμε τους απασχολούμενους, για να αποφύγουμε, πώς να το πω, την επικάλυψη ή τον τριπλασιασμό των περιπτώσεων στο, αυτών στο δρόμο, γιατί το μόνο που μπορούν να συνεπάγονται είναι επιδείνωση των συνθήκων ε, των μεταφορών. Οπότε για την οδική ασφάλεια μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αναγνωρίζει πως μπορεί να ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση, αλλά χρειάζεται μεταβατική περίοδος. Μάλιστα. Η, η οδηγία μέχρι το 2009 ε, θα παρέμενε σε ισχύ και είμαστε τώρα στο 2009. Οπότε η υπόσχεση της Επιτροπής ήταν να εφαρμοστεί η οδηγία σε όλους τους οδικούς μεταφορείς, μισθωτούς και αυταπασχολούμενους. Και υπάρχουν εδώ στην αίθουσα και άλλοι βουλευτές που ήταν μαζί μου σε εκείνη τη συζήτηση στην Επιτροπή. Μα αυτό μας είχε υποσχεθεί η Επιτροπή, ότι από το 2009 και μετά έπρεπε να εφαρμοστεί η οδηγία σε όλους. Και το χρόνο πρέπει να τεθεί σε ισχύ αυτό, υπαναχωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τι κάνει, υποβάλλει νέα πρόταση για να εμποδίσει την εφαρμογή της διάταξης σε όλους. Και για να επιστρέψουμε στην πρώτερη κατάσταση. Ενώ μας είχε υποσχεθεί το 2002, το 2009 θα ρυθμιζόταν η κατάσταση. Και ξαφνιάζομαι γιατί συζητάμε εδώ τώρα για την δυνατότητα σύναψης ε, συμφωνιών. Ε, λέμε να ξανανοίξουμε το φάκελο, θέλουμε να δούμε τις προϋποθέσεις, αλλά ο εκπρόσωπος της Επιτροπής τα ίδια επιχειρήματα μας σερβίρει. Τα ίδια που ακούσαμε το Μάιο τότε, το 2002. Και Κανένα μήνυμα δεν μας περνάει ότι είναι ανοιχτός ε, σε αυτή την ε, δυνατότητα εφαρμογής ε, της οδηγίας σε όλους, όλους τους Δεν Μιλάμε για μισθωτούς, για αυτοαπασχολούμενους, ψευδοαπασχολούμενους και ούτω καθεξής. Ναι, ναι, Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω. Εγώ πιστεύω πως η Επιτροπή μας ε, τοποθετείται σαφώς ε, σε αυτό το θέμα και πρέπει να εμείνουμε στην θέση που εγκρίναμε εκείνο το Μάιο στο Κοινοβούλιο. Και... Η θέση του Μαΐου συνάδει με τη θέση του 2002. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Μίλαν Τσαμπνό και κυρία Σαρή Σαγιά. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, na okraji uvádím, že mě mrzí, že naše frakce nedostala možnost vystoupit v rámci... Ευχαριστώ κυρία Δεν ζητήσατε να μιλήσει κανεί και ο όδησης από την πολιτική μου ομάδα. Ελπίζω να μην κάνετε το ίδιο λάθο την επόμενη φορά. Ε, Τέλο πάντων, επί του προκειμένου. Ε, Υπάρχει η οδηγία του 2002, ε, βελτιώθηκαν ορισμένα πράγματα, αλλά εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ε, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει ανάγκη να ε, νομοθετήσουμε περαιτέρω γιατί δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να νομοθετήσουμε τους αυτοαπασχολούμενους δεν είναι υπάλληλο κάποιου αυτοαπασχολούμενος παίρνει τις αποφάσεις του μόνος του και υπάρχουν από εκεί και πέρα για την οδική ασφάλεια οι οδηγίες του 2006-2005 υπάρχουν συνθήκες και ε, φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα με τη γερμανική μετάφραση. La cabine allemande est rétablie? Aha, sorry, I didn't know that. Sorry. C'est rétabli? Yeah. Bon, très bien. Merci de. May I repeat it? Euh, euh, pouvez conclure en une phrase. Μπορείτε να επανα... μια φράση να πείτε μονάχα για να τελειώ. Λοιπόν, εγώ λέω ότι δίκιο έχει κυρία Edith Bauer. Θέλουμε νέα έκθεση. Ωραία, ευχαριστώ. Σαρία Σαγιά και μετά κυρία Λαμπέχ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την αναζήτηση για κάποια συμβιβαστική λύση. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου δεν γίνεται κανένας έλεγχος και δεν εποπτεύεται η εφαρμογή των νομοθετικών πράξεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ε, οι αυτοαπασχολούμενοι δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στην οδηγία. Και από άποψη οδικής ασφάλειας οι κανόνες για, τους, χρόνου το χρόνο οδήγησης και χρόνο ανάπαυσης είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Αν, αν κατάλαβα καλά, κάποιοι συνάδελφοι εδώ είπαν ότι δεν χρειάζεται καν ε, να τεθούν κανόνες για την, το χρόνο οδήγησης και χρόνο ανάπαυσης και βεβαίως το μπορούμε να ελέγξουμε τι κάνουν ε, οι άνθρωποι στο χρόνο ανάπαυσή του. Μπορούν να πάνε να δουν τηλεόραση, μπορούν να κοιμηθούν, μπορούν όμω να πάνε σε πάρτι, να πιούνε, να καπνίσουν κλπ. το να βλέπουμε λοιπόν, το να έχουμε κανόνε για το τι κάνει ο άλλο στο χρόνο ε, ανάπαυσή του είναι εξωφρενικό. Αλλά μπορούμε να, παρα, να δούμε τι γίνεται ε, κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας στη Φινλανδία μια πρόσφατη μελέτη ε, είδαμε ότι τρία τέταρτα των ε, ε, θυμάτων, των ατυχημάτων ε, οφείλονταν σε κάτι τι άλλο εκτός από την οδήγηση αυτή καθεαυτή τι περισσότερες φορές ε, έφταιγαν οι δρόμοι, οι ολιστηροί δρόμοι, κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν οι οδηγοί κτλ. Κυρία Λαμπέρ, ευχαριστώ πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω στα θέματα τη τα διαδικαστικά αν θέλετε, όχι σε θέματα ουσία. Ρωτώ λοιπόν, οι νέε συζητήσει που λαμβάνουν χώρα, και για τις οποίες μας μίλησαν είναι επί της ουσίας ή είναι της διαδικασίας και σχετικά με την ψηφοφορία που έλαβε χώρο στο Κοινοβούλιο. Γιατί εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο με βάση την τωρινή πρόταση που υπάρχει να βρω οποιαδήποτε συμβαστική ε, λύση και μετά από την παρέμβαση και της Κομισιόν σήμερα το απόγευμα θεωρώ ότι είμαστε διαμετρικά αντίθετοι οι με τους δε και άρα δεν βλέπω να υπάρχει ενδεχόμενο συμβαστικής λύσης. Εγώ νομίζω ότι αν δεν γίνουν επίσημες ουσιαστικές συζητήσεις δεν πρόκειται να βγούμε από το αδιέξοδο. Άρα αξίζει, ε, βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι οι συζητήσει που κάνουμε δεδομένε τη θέση τη Κομισιόν όπω είπα προηγουμένω, ε, δεν θα αποδώσουν ε, καρπού. Ε, μακάρι να βρίσκαμε συμβαστική λύση αλλά νομίζω πως δεν θα βρούμε. Γι' αυτό πρέπει να γίνει νέα έξεση τελικώς. Πασκάλ Γκρουνιέ και μετά κύριο Στούσας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ σπάνια είμαι υπέρ των περιορισμών για το χρόνο εργασίας, αλλά εφόσον μιλάμε για την οδήγηση, ε, αλλάζει το πράγμα και δεν καταλαβαίνω γιατί ε, πρέπει να αποκλειστούν οι αυτοαπασχολούμενοι από την οδηγία για το χρόνο εργασίας. Εάν ε, ε, μιλάμε για την οδική ασφάλεια και δεν θέλω να ξαναρχίσω τώρα τη συζήτηση και να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, απλά θέλω να σας πω ότι στη Γαλλία έχουμε πολύ λιγότερα ατυχήματα που εμπλέκονται φορτηγά, αλλά αν αληθεύει αυτό, αληθεύει για την τελευταία δεκαετία και οφείλεται στο ότι ρυθμίσαν πολύ καλά το χρόνο εργασίας για του μισθωτού. Γιατί εμεί έχουμε πολλού οδηγού που είναι μισθωτοί και άρα τα μέτρα είχαν πολύ σημαντική επίπτωση στη μείωση και οδήγησαν σε μεγάλη μείωση των ατυχημάτων. Αλλά εμένα με ενοχλεί ο στρεβλωμένο αθέμητο ε, ανταγωνισμό. Δηλαδή να ζητάνε οι εταιρείε από, τις, από το τους εργαζόμενους τους για να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι, για να παρακάμψουν την οδηγία. Ε, αυτό μπορεί να συμβεί σε όλα τα κράτη-μέλη και εφόσον είναι εντελώ διαφορετική ε, η νομοθεσία, εμεί είμαστε χώρα διαμετακόμιση και άρα έχουμε πρόβλημα με τον αθέμητο ανταγωνισμό. Και θα ήθελα να το ληφθεί υπόψη τώρα για την εξακρίβωση για τον έλεγχο, ναι, δύσκολο είναι. Πώ να ελέγξει κανεί τον χρόνο εργασία των αυτοαπασχολούμενων. Εγώ έχω μια επαγγελματική εμπειρία στι μεταφορέ, ξέρετε, και μπορώ να σα πω ότι μπορούμε. ότι πέρα από τον ταχυγράφο έχουμε και τους χρόνους φόρτωσης ε, εκφόρτωσης. Ε, πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη για να ξέρουμε ποιος είναι ελάχιστος και ο τους χρονος εργασίας ε, Ήδη από το Μάρτιο 2009 κατά αυτόν τον τρόπο έπρεπε να έχει εφαρμοστεί η οδηγία. Μάλιστα σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Τούσας και ο κύριος Έτσο Κομφεράτη. Κύριε Τούσα. Με θεσμοθετημένες 84 ώρες δουλειά τη βδομάδα για τους εργαζόμενους στις κοινικέ δραστηριότητες των οδικών μεταφορών και σε συνδυασμό με τους ψευδοαπασχολούμενους και τους αυτοαπασχολούμενους δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στην οδική ασφάλεια και αυτό είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο. Παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή την ομιλία εκ μέρους της Επιτροπής. Είναι ανυπόστατη η ισχυρισμή και τα επιχειρήματά τους. Και επιπρόσθετα προηγούμενη ομιλήτρια έθεσε το θέμα το ότι είχαν δεσμευτεί για την εφαρμογή της νομοθεσίας τόσο σε ό,τι αφορά για το 2009, τόσο σε ό,τι αφορά για τους μισθωτούς, όσο και για τους αυτοαπασχολούμενους. Δεν είναι σωστό ότι να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία για μια νέα συμφωνία, για μια νέα πρόταση, γιατί αλλιώς δεν συμφέρει σε τίποτα. Ίσα ίσα μια τέτοια κατέθεση και πρόταση θα οξύνει τα προβλήματα και τα αποτελέσματα θα είναι οδυνηρά τόσο για τους ίδιους τους οδηγούς των αυτοκινήτων αλλά και όλους όσους χρησιμοποιούμε τους οδικούς άξονες. Και τέλος πάντων, ας είμαστε καθαροί μεταξύ μας. Αυτούς που εξυπηρετεί είναι τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που βρίσκουν διάφορους τρόπους να χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους. Αν θέλουμε να πάρουμε μέτρα και χρειάζεται να πάρουμε μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να το δούμε και σε άλλο, σε άλλο επίπεδο και να δούμε πώς θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα κεφαλαιόδε ζήτημα που έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια. Οδική ασφάλεια και γι' αυτό πρέπει άμεσα να πάρθει ε, μέτρα και γι' αυτό το τομέα. Νομίζω ότι αύριο πρέπει κανονικά να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ο κύριος Σερτζό Καμφεράτη και μετά ο κύριος Σωρή. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν μια πολύ σύντομη ερώτηση ως προς τη μέθοδο. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να συζητήσουμε. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει από τότε που ψήφισε το Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχουν επιχειρήματα τα οποία ε, μας δίνουν ε, λόγους για να ξανασυζητήσουμε ένα θέμα. Να περάσω τώρα στην ουσία. Τα προβλήματα που αφορούν στα οδικά ατυχήματα, η έλλειψη ασφάλειας στους δρόμους έχουν τρεις συνιστώσεις την κατάσταση των ε, αυτοκινήτων οχημάτων, την κατάσταση των ε, οδικών αξώνων και την κούραση των οδηγών. Η κούραση σχετίζεται με τον ποσότητα εργασία, τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουν την εργασία του και τι ώρε που δουλεύουν. Ανεξάρτητα από το αν είναι εργο, εργαζόμενοι ή αν είναι αυτοαποσχολούμενοι, δεν φαντάζομαι να υπάρχει άλλο μέρος του κόσμου που γίνεται αυτή η διάκριση. Αν υπάρχει ένας κανόνας και εισάγεται ένα του κανόνας, σαφώς υπάρχει κάποιος κόστος. Αν υπαρχει ενα κανονα και εισαγεται ενα κανονα σαφω υπαρχει καποιο κοστο αν λοιπον λοιπόν δεν εφαρμοστεί συνολικά υπάρχουν δύο πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Αυξάνεται ο ανταγωνισμός και ε, αλλάζουν τα δικαιώματα των ατόμων. Τα άτομα τα οποία εργάζονται ε, έχουν κάποια δικαιώματα τα οποία θα διασφαλίζουν και τη δική τους την ασφάλεια και δεν θα πρέπει να τα στερούνται κάποιοι πολίτες. Αν υπάρχουν κανόνες που κάνουν διάκριση χωρίς να υπάρχει λόγος έναν ε, τομέα, ε, θα πρέπει να υπάρχει αλλαγή, αλλιώς ευνοούνται η παρέκκληση, η απομάκρυνση από τον αρχικό κανόνα και τελικά θα καταλήξουμε σε κάποιες περιπτώσεις οι οποίες ε, θα ε, είναι στρεβλωμένες σε σχέση με τις αρχικές καταστάσεις. Αναφέρω κάτι τελευταίο, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι η δυνατότητα να δώσουμε ίσως στα κράτη-μέλη ε, να κάνουν κάποιες ε, παρεκκλήσεις από τους κανόνες. Λέτε ότι αυτά γίνονται κατά ε, προέκταση. Αλλά αν τα πράγματα έχουν εκεί, ποιο είναι ένα κράτος, το κράτος το οποίο θα αυξήσει το κόστος σε κάτι. Επίσης, μιλάμε για δραστηριότητες οι οποίες ούτως ή άλλως αφαιρούν εδώ και αρκετό καιρό την όλη ευρωπαϊκή επικράτεια. αν δεν έχουμε τη δυνατότητα επέκτησης, ουσιαστικά ε, αρνούμαστε την ίδια την Ευρώπη. Επιτρέπουμε σε κάποιους να έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και δεν θα έχουμε μόνο κοινωνικό ντάμπινγκ, αλλά θα έχουμε και κοινωνικό ε, ντάμπινγκ. Ο κύριος Σωρή, ε, ζητώ συγγνώμη, έχετε ζητήσει το λόγο εδώ και αρκετή ώρα, αλλά δεν σας είδα. Και μετά ο κύριος Διτερκό που θα είναι τελευταίος πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Ο κύριος Σωρή. Εκτός μικροφώνου μιλητής. εγώ ναι. Να έχω έναν οδηγό που ε, να βρεθώ αντιμέτωπος με έναν οδηγό ο οποίος οδηγούσε 20 ώρες και πριν οδηγήσει 20 ώρες είχε κάνει και κάτι ακόμα. Θεωρώ λοιπόν ότι ο χρόνος οδήγησης θα πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρός και να ρυθμίζεται με τους χρονοταχυγράφους. Τώρα, το Επιτροπή να ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση και για τα 27 κράτη-μέλη. Ξεκινάμε λοιπόν μια θεσμική διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπώνησαν μια νομοθεσία που τα κράτη-μέλη απλώς δεν θέλουν να την εφαρμόσουν. Αυτό λοιπόν με κάνει να αναρωτιέμαι. Αξίζει ο κόπος να σκεφτούμε ένα συμβιβασμό για μια τέτοια μορφή νομοθεσία. θα πρέπει να σκεφτούμε και τους εργαζόμενους, διότι οι εργαζόμενοι δεν αποφασίζουν αυτόνομα πώς θα οργανώσουν το χρόνο εργασίας τους, επομένως δεν θα πρέπει να δημιουργούμε διακρίσεις. Είναι αλήθεια ότι το Κοινοβούλιο πήρε μία απόφαση με μία οριακή πλειοψηφία Κατά την άποψή μου όμως δεν θα πρέπει ε, να εμένουμε σε αυτές τις θέσεις. Υπάρχουν προσκόμματα, ε, αλλά θα μπορούσε ίσως το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουν κάτι για να βελτιώσουν οι ίδιοι αυτή την πρόταση. Θα ακούσουμε τον κύριο Ντίτερκο που είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ε, Κύριε Ωρή, Είπα στην αρχή τη συζήτηση ότι το Συμβούλιο μα είπε ότι μα εμπιστεύεται, εμπιστεύεται τη σοφία του Κοινοβουλίου. Τι να κάνω εγώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. τρει ε, παρατηρήσει πρωτα Πρώτα-πρώτα, για όλου πρέπει να ισχύουν οι χρόνοι οδήγηση και ανάπαυση Δεύτερα, θεωρώ ε, φοβερό λάθος και παραπλανητικό αν θέλετε ε, το να κάνουμε διάκριση μεταξύ αυτοαποσχολούμενων και μη. Είναι αδύνατο αυτό. Ε, και τρίτον, αυτοί οι οποίοι φωνάζουν για την οδική ασφάλεια θα πρέπει, είναι μη συνεπείς. Γιατί θα έπρεπε να πούμε όποιος έχει δουλέψει 8 ώρα δεν μπορεί να επιτρέπεται να οδηγεί, να μπαίνει στο αυτοκίνητο να οδηγεί. Δεν το θέλω εγώ αυτό. Ε, ε, λοιπόν, μπορείτε να μας διαφωτίσετε για την ε, στρατηγική που προτείνετε. Τι ακριβώς δηλαδή μπορούμε να αποφασίσουμε. Köszönöm Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Πιστεύω ότι είναι ψευδές να πούμε ότι η οδική ασφάλεια είναι ένα θέμα που θα ρυθμιστεί με αυτό το κείμενο. 561 του 2004 αφορά στην οδική ασφάλεια. Κάτι που μπορούμε να μάθουμε από αυτή τη συζήτηση είναι ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με τους ψευδοαπασχολούμενους. Για να έχουμε ένα θεμητό ανταγωνισμό, πρέπει να δεχτούμε τους ίδιους κανόνες ε, για όλους, είτε πρόκειται για αυτοαπασχολούμενου ή ψευδοαπασχολούμενου, και δεν μιλώ εδώ μόνο για τις οδικέ ε, μεταφορές, μιλώ για ολόκληρη την οικονομία. Αν θέλουμε να συζητήσουμε το θέμα των ε, ψευδοαπασχολουμένων μόνο, ας κάνουμε ξεχωριστή έκθεση, ας κάνουμε έκθεση πρωτοβουλίας. Υπάρχει ε, το πρόβλημα και καλούμαστε να το λύσουμε. αν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα που σχετίζονται με του ψευδοαπασχολούμενου, χρειαζόμαστε ξεχωριστή έκθεση. Δεν μπορούμε να προσπαθούμε μέσα από αυτό το κείμενο να λύσουμε τα προβλήματα που σχετίζονται με του ε, ψευδοαπασχολούμενου. Ο χρόνο εργασία των αυτοαπασχολούμενων είναι αδύνατον ε, να ελέγχθει. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά χρήματα και απεριόριστο χρόνο για να ελέγξουμε το χρόνο εργασία των αυτοαπασχολούμενων. Ε, με ρωτήσατε ποιες λύσεις μπορώ να προτείνω, ποιες στρατηγική μπορώ να προτείνω. Θα σας ζητήσω λίγο περισσότερο χρόνο για να ακούσω και τις απόψει των κοινωνικών εταίρων. Ήδη ε, είχαμε κάποιες επαφές. Καλό είναι πάντοτε να ακούμε τις απόψεις των άλλων και να μην λέμε ότι εμείς είμαστε οι πιο ευφυείς και εμείς είμαστε πλέον αρμόδιοι για να ρυθμίσουμε το ζήτημα. Το Συμβουλίο και η Επιτροπή έχουν ε, επίσης οργανώσει διαβουλεύσει. Πρέπει να ακουστεί άποψη όλων πριν αποφασίσουμε. Θα ήθελα να σας ζητήσω να ξαναδώσετε το θέμα στους συντονιστές για να αποφασίσουν αν τελικά θα συντάξουμε άλλη έκθεση ή αν θα ψηφίσουμε για αυτήν την έκθεση. Κάποιοι συνάδελφοι ζήτησαν νέα έκθεση. Άλλοι πάλι ε, πιστεύουν ότι πρέπει να ψηφίσουμε για αυτήν την έκθεση. Ε, πλεονεκτήματα και μενεκτήματα υπάρχουν και στις δύο περιπτώσεις. Σας ζητώ, Πρόεδρε, να ε, δώσετε την απόφαση, να αφήσετε τους συντονιστές να πάρουν την απόφαση, η Πρόεδρος. Ε, μάλιστα, ευχαριστούμε. Εγώ θα σας κάνω μια ελαφρώς διαφορετική πρόταση μπορούμε να ελέγξουμε και τι έγινε στα πρακτικά της Ολομέλειας ε, για να θυμηθούμε τις συνθήκες ε, υπό τις οποίες ε, αναπέμφθηκε η έκθεση στην Επιτροπή μας επί τη βάση του παλιού 52,3 που τώρα είναι το 56,3 και μας επιβεβαιώνει είτε να επιβεβαιώσουμε τη θέση είτε να υποβάλουμε νέα έκθεση αναπέμφθηκε στην Επιτροπή μας και όχι στους συντονιστές της Επιτροπής μας δεδομένου, όμως το δεδομένες της πλούσιας συζήτησης που μόλις έγινε, θεωρώ ότι ακούσαμε, εκφράστηκαν όλες οι απόψεις και άρα στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας, δηλαδή στις 29 Σεπτεμβρίου, προτείνω να ψηφίσουμε για την έκθεσή σας. Ανάλογα με την έκβαση της ψηφοφορίας, είτε θα επιβεβαιωθεί η θέση και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια, δηλαδή την πρόταση απόρριψη τη πρώτα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε δεν θα επιβεβαιωθεί η θέση από τη νέα Επιτροπή Απασχόληση με τη νέα σύνθεσή τη και εν τη αυτή περιπτώση επαφίεται σε εμά ή στου συντονιστέ να αποφασίσουν ποιο πρέπει να εκπονήσει νέα έκθεση. Συμφωνείτε? Υπάρχουν στάσει για ε, αυτή τη ε, διαδικασία που σα προτείνω. Για να το πω σαφέστερα, ε, στις 29 Σεπτεμβρίου, στην επόμενη συνεδρία, θα ψηφίσουμε για την έκθεση της κυρίας Μπάουερ ως έχει. Και αν επιβεβαιώσουμε την έκθεση της κυρίας Μπάουερ, αυτό σημαίνει ότι προτείνουμε στην Ολομέλεια να διατηρήσει τη θέση της, δηλαδή να συνεχίσει να απορρίπτει τη θέση της Επιτροπής. Ή αν απορριφθεί από εμά η έκθεση, θα πρέπει να εκπονηθεί νέα έκθεση. Ε, μπορούμε να κλείσουμε με αυτό το συμπέρασμα τη συζήτησή μας. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό θα κάνουμε. Το σημείο 6 αύριο θα το δούμε. Ε, ζητώ συγγνώμη από τους προσκεκλημένους μας. Με πάσα ειλικρίνεια, αλλά καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ήταν το θέμα που συζητούσαμε. Κύριε Έρη, διαδικαστικό. Πρόεδρε, εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα. Ε, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, δεν νομίζω να σημειωθεί πρόοδος. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα στους συντονιστές, να ληφθεί η απόφαση από τους συντονιστές. Αν ε, ανέκαθεν αυτό κάναμε. Είναι μια παράδοση, έτσι. Ε, εκείνοι αποφασίζουν. Μα όχι, δεν έχουν εξουσία να επιβεβαιώνουν, να κυρώνουν θέση της Επιτροπής Συντονιστές θα κάνουμε αυτό που είπα εφόσον συμφώνησε η εισηγήτρια και τα μέλη της Επιτροπής. Ζητώ συγγνώμη όπως έλεγα από τους προσκεκλημένους μας. Ε, τους ευχαριστώ για την παρουσία τους. Ζητώ, παρακαλώ όλους όσους φεύγουν από την αίθουσα να το κάνουν ε, σιωπηρά, χωρίς θόρυβο. Και ζητώ από τον κύριο Ροντρίγκες, από την Ένωση ΝΤΑΣ, και από τον Κλοντ Μανιουέλ Τριόμφ από την Άστρε. Έχετε αποφασίσει μάλλον εσείς με ποια σειρά θα κάνετε τις παρουσιάσεις. Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε ε, για την ε, μελέτη, για τον αντίκτυπο των νέων μορφών εργασία βιομηχανικές βιομηχανικέ σχέσει και στην εξέλιξη τη εργασιακή νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγο περαιτέρω καθυστέρηση. Πείτε μα απλώ ποιο μιλάει. Και θα σας ακούσουμε με ιδιαίτερη προσοχή παρακαλώ και πάλι μην κάνετε θόρυβο όσοι φεύγετε από την αίθουσα. Σας παρακαλώ. Ησυχία. Ε, ο κύριος Δροντρίκης ή ο κύριος Τρεόμφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν χαρά μου που παρακολούθησα τη συνεδρίασή σας. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον για μας. Κάποια από τα θέματα άλλωστε που συζητήθηκαν ε, προηγουμένως εδώ είναι πολύ ενδιαφέροντα και ε, έχουν να κάνουν και με τη μελέτη μας. Είναι πολύ δύσκολο να συνοψίσουμε σε 10 λεπτά τα όσα έχουμε κάνει το 2007 και το 2008, αλλά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό κάνουμε από κοινού αυτή την παρουσίαση με τον συνάδελφο. Προσπαθήσαμε να επικαιροποιήσουμε λίγο τα αποτελέσματα της μελέτης μας και να συμπεριλάβουμε και κάποιες αναφορές, κάποιες σκέψεις για την ε, υφιστάμενη κρίση, διότι η ε, μελέτη μας όπως σας είπα έγινε στην αρχή της κρίσης, στις αρχές του 2008, επομένως Να δούμε λίγο την επόμενη διαφάνεια. Αυτά που κάναμε λοιπόν ήταν ουσιαστικά να δώσουμε μια συνοπτική εικόνα των βασικών χαρακτηριστικών και των ε, ε, τρόπων που γίνονται οι συμβάσεις στα 27 κράτη-μέλη. Έχουμε λοιπόν τη δέσμευση που αναλάβαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιμετωπίσουμε τα θέματα τα οποία προέκυψαν από την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εξυγχρονισμό, τον τρόπο εργασίας και τις προκλήσεις που έχουμε στον 21ο αιώνα και να λάβουμε υπόψη μας και τις επιπτώσεις της ε, άτυπης εργασίας ε, και την, ε, να μπορέσουμε να τα συμπεριλάβουμε αυτά και στο εργασιακό δίκαιο. Σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή τη μελέτη, αναλύσαμε επίσης και τις επιπτώσεις ε, του εργατικού δικαίου όχι μόνο ε, βασιζόμενο στις σχέσεις που έχουμε μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενο αλλά και στον κοινωνικό διάλογο και στις οικονομικές συνέπειες. Κάναμε μια ανάλυση της αγοράς εργασίας, της εξέλιξης της αγοράς εργασίας ε, στα 27 κράτη-μέλη, λαμβάνοντας υπόψη και νέους ε, τρόπους εργασίας. Επίσης, ε, χρησιμοποίησαμε και τρεις ε, περιπτωσιολογικές μελέτες, οι οποίες αφορούν σε διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, ε, κυρίως για τις συμβάσεις εργασίας, θέματα flexicurity, ευελικτή και ποια είναι τα συμπεράσματά μας εν συντομία στην επόμενη διαφάνεια. Καταρχάς, βρήκαμε πάρα πολλές διαφορετικές μορφές ε, εργασίας, ακόμα περισσότερες από αυτές που περιμέναμε. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι ότι πολλές μορφές εργασίας συμπεριλαμβάνονται στις μελέτες μας, έχετε αυτή τη μελέτη ε, στη διάθεσή σας, αλλά διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές νέες μορφές ε, άτυπων συμβάσεων εργασίας. Διαπιστώσαμε επίσης ότι όντως αυτές οι νέες μορφές εργασίας αυξάνονται συνεχώς. Ε, έχουμε δεδομένα ε, στατιστικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από προσωπικές αξιολογήσεις και από ε, την προσωπική μας ανάλυση της αγοράς εργασίας και καταδεικνύεται σαφώς αυτό το φαινόμενο. Τρίτον, διαπιστώσαμε ότι αυτές οι διαφορετικές μορφές εργασίας ε, λαμβάνονται υπόψη με διαφορετικό τρόπο. Προσπαθήσαμε να καθορίσουμε τρεις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη είναι η άτυπη σχέση εργασίας και εδώ διαπιστώνουμε ότι έχουμε και ε, προσωρινή εργασία, ε, εργασία μερική απασχόληση, ε, αυτές οι σχέσεις εργασίας διαφέρουν από τις συνήθεις σχέσεις εργασίας, την πλήρη απασχόληση, ε, την σύμβαση αορίστου χρόνου και ούτω καθεξής. Μια άλλη κατηγορία είναι ε, οι ειδικέ ε, σχέσεις μη απασχόλησης, μιλάμε για αυτοαπασχόληση δηλαδή και οικονομικά ανεξάρτητη εργασία, ε, καθώς επίσης και νέες μορφές τριγωνικών σχέσεων πέρα από τις ε, θέσεις προσωρινή απασχόληση. Έχουμε υπερβο... οι σχέσεις υπεργολαβίας, για παράδειγμα, μεταξύ επιχειρήσεων και υπάρχει και μια τρίτη βασική κατηγορία που είναι οι, άδε... οι άλλες μορφές εργασίας οι οποίες δεν ρυθμίζονται σωστά. Παραδείγματος χάρη τηλεεργασία, εκπαίδευση, ε, πολλές διαφορετικές μορφές εργασιακών σχέσεων. Κάποιες από αυτές ε, θεωρούνται άτυπες θέσεις εργασίας σε κάποιες χώρες, αλλά ρυθμίζονται ως σχέσεις μη εργασιακές σε κάποιες άλλες χώρες. What about the impact on labor law and Οι επιπτώσεις λοιπόν στο εργατικό δίκαιο και στις αγορές εργασίας διαπιστώσαμε ότι η έννοια της ε, σχέσης απασχόλησης θα πρέπει να επανεξεταστεί. Θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω εδώ ότι υπάρχει μία σύσταση του 1998 και εγκρίθηκε από εκεί και πέρα το 2006 για τις σχέσεις εργασίας. Εγκρίθηκε και από τα κράτη-μέλη Σχεδόν με μεμοφωνία είχαμε δύο αποχές και το, το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακίνησε τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τη σύσταση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας του 1998. Αυτές οι νέες μορφές εργασίας, οι οποίες έχουν προκύψει, έχουν διάφορες μορφές άτυπης εργασίας και όλες αυτές έχουν όλο ένα και αυξανόμενες περίπλοκες νομικές μορφές εργασίας. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αυτές οι νέες μορφές ε, εργασίας, διότι συνεισφέρουν και στην, ε, στην στον κατακαιρματισμό της ε, αργόρας εργασίας και όλα τα κράτη-μέλη πλήττονται από αυτό το φαινόμενο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το εργατικό δίκαιο και οι κοινωνικές ασφαλίσεις έχουν βασιστεί στις βασικές παραδοσιακές μορφές εργασίας, δηλαδή την πλήρη απασχόληση και τις συμβάσεις αορίστου χρόνου. Ε, συνήθως ε, ε, λαμβάνουμε υπόψη αυτή τη μορφή προστασίας κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, υπάρχουν ε, μία σειρά από εργαζόμενοι που καταδεικνύουν διαφορετικά χαρακτηριστικά εργασίας ταυτόχρονα. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, εργαζόμενοι που μπορεί να έχουν σύμβαση εργασίας και ταυτόχρονα να εργάζονται με μερική απασχόληση και κάπου αλλού. Κάτι ακόμα το οποίο θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε είναι τα συλλογικά δικαιώματα. Ήταν πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε μια κοινή τάση στα κράτη-μέλη για τις επιπτώσεις ε, των αλλαγών ε, που σας επεσήμανα στα συλλογικά δικαιώματα. Έχουν να κάνουν με τα ε, συστήματα εργασίας σε κάθε χώρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό της. Ε, εκείνο που είναι αλήθεια είναι ότι διαπιστώσαμε ότι μπορεί να επηρεαστούν και να περιοριστούν τα συλλογικά δικαιώματα λόγω το γεγονότος ότι τα περισσότερα ε, εργασιακά δικαιώματα έχουν εγκριθεί ε, βάσει ενός μοντέλου σύμβασης αορίστου χρόνου. Και θα πρέπει να το εξυγχρονίσουμε λίγο αυτό. Τώρα, ο κοινωνικός διάλογος και οι συμφωνίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο νομίζω ότι διαδραματίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και λόγω διάδοσης και λόγω προσαρμονικής της χρήσης των ε, συμβατικών μορφών μέσω ε, εσωτερικής ευελιξίας. Υπάρχουν λοιπόν συμφωνίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, οι οποίες έχουν υπάρξει αντικείμενο συμφωνίας από τους κοινωνικούς εταίρους και συνεισφέρουν και ανοίγουν το δρόμο για την εφαρμογή αυτών των νέων μορφών εργασίας. Τέλος, έχουμε δεν έχουμε, συγγνώμη, ενδείξεις ε, για το ρόλο της ήπιας νομοθεσίας, του soft law. Δεν φαίνεται να αντικαθιστά το παραδοσιακό εργασιακό δίκαιο. Φαίνεται ότι στην πλειονότητα των κρατών μελών ε, το εργασιακό δίκαιο ε, εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αντίθεση με το ενήπια νομοθεσία. Ε, αλλά υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για την ανάπτυξη εταιρικής κοινωνικής ε, ε, ευθύνης, κώδικες διοντολογίας σε κάποιες χώρες, σε κάποια συστήματα φαίνεται να διαδραματίζουν ολαιόνα και σημαντικότερο ρόλο αυτά τα στοιχεία. Εδώ τώρα Έχουμε την επόμενη διαφάνεια. Μας ρωτήσατε και για το ρόλο της ευελικτασφάλειας, του flexicurity στα τελευταία χρόνια, τις επιπτώσεις στο εργασιακό δίκαιο και τις επιπτώσεις ε, στα ε, συστήματα εργασίας. Η προσέγγιση της ευελικτασφάλειας δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι ένας τρόπος για να επιτύχουμε το στόχο ε, του να έχουμε περισσότερη ευελιξία, να έχουμε περισσότερη ανταγωνιστικότητα, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και ασφάλεια που σχετίζεται με το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Είναι αλήθεια ότι καταρχάς η flexicurity συμπεριλαμβάνεται σε κάποιες από τις βασικές ε, κατευθυντήριες γραμμές για την στρατηγική για την απασχόληση. Στα τέλη του 2007 εγκρίθηκε στο Συμβούλιο και όλο ένα και περισσότερο αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο με διάφορες μορφές ε, μέτρων για την ευελικτή ασφάλεια. Το πρόβλημα είναι και ότι το θέμα αυτό είναι διαφιλονικούμενο στα περισσότερα κράτη-μέλη αν ε, ρωτήσουμε τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά ακόμα και ακαδημαϊκούς, διότι φαίνεται, ναι μεν οι βασικές αρχές της ευελικτασφάλειας καλύπτουν τα πάντα, αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά καταλήλως. Και διαπιστώσαμε θα πρέπει λοιπόν η εφαρμογή της θα πρέπει να βασίζεται σε συμπεφωνημένο κοινωνικό διάλογο και να δούμε πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε καταλήλως τις επιπτώσεις. Σε, κάποιες κράτη, σε κάποια κράτη-μέλη έχει συζητηθεί ε, ίσως και η ύπαρξη κάποιων ανεξαρτήτων φορέων που θα μπορούσαν να αναλάβουν την παρακολούθηση, την εποπτεία και να δούνε ότι έχουμε μια καλά ισορροπημένη προσέγγιση και μια καλή προσαρμογή στη flexicurity. Βεβαίως, καλή ισορροπία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Είδαμε ότι πραγματικά εφαρμόζουν τις αρχές Flex Security κάποια κράτη-μέλη πολύ εξισορροπημένα. Αλλά εφαρμόζουν τα, τις αρχές Flex Security ως άλοφη για να κάνουν άλλα πράγματα. Βεβαίως όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να ε, εφαρμόστα προσαρμοστούν στην ε, παράδοση και στην κουλτούρα της χώρας στην οποία εφαρμόζεται. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τα ίδια πράγματα ε, μέσα στην εργασιακή κουλτούρα της Δανίας και της Ολλανδίας όπως στο νότο της Ευρώπης παραδείγματος χάρη. Εν πάση περιπτώσει ε, επίσης θα πρέπει η εφαρμογή της flexicurity να στηρίζεται από δημόσια, δημόσιους πόρους για να μπορέσουν να ε, βοηθηθούν ε, οι οποιασδήποτε εργασιακές μετατροπές ε, χρειάζεται να, γίνουν. Βεβαίως η οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή επιβάλλει λιτότητα και περιορισμού στους εθνικούς προπολογισμού, οπότε αυτό το τελευταίο είναι δύσκολο. Θα μιλήσω γαλλικά και θα σας πω ποια είναι τα συμπεράσματα της μελέτης μας. Δυο είναι τα σημαντικά συμπεράσματα. Πρώτα πρώτα να αρχίσουμε αλλιώ. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που απορρέουν από τούτη εδώ την μελέτη. Θα μπορούσαμε να τα κατηγοριοποιήσουμε γύρω από τέσσερις άξονες, τέσσερα σημεία. Πρώτο, προσαρμογή σε, στη, παρόλο που γίνονται προσαρμογές ε, ανάλογα με τους νέους τύπους εργασίας ε, δυστυχώς αυτό δεν εξασφαλίζει ισότητα. Δηλαδή βλέπουμε de facto, αν όχι de jure, ανισομέρειες εφαρμογής. Οι νέες μορφές εργασίας, οι άτυπες μορφές εργασίας δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά για να μπορούν να ανταποκριθούν στην ανάγκη για ε, δικαιοσύνη και ίση μεταχείριση. Είναι αν οι ανισομέρειες, οι ανισότητες είναι τεράστιες ιδιαίτερα σε σχέση με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για τις νέες μορφές εργασίας. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, ε, τα αλλαγή αν θέλετε ή τα αλλαγή ε, κατεύθυνση των εργαζομένων εάν και εφόσον ε, κλείσει η επιχείρηση ή κάνει μια κάποια αναδιάρθρωση κτλ. Ε, ωραία. Αυτά όλα δεν γίνονται με ίσο τρόπο, με ίδιο τρόπο για όλους, ούτε de facto ούτε de jure. Τρίτο θέμα. Η ίδια συμμετοχή σήμερα αυτών των εργαζομένων των νέων μοφών εργασίας δηλαδή στον κοινωνικό διάλογο είναι πολύ διαφορετική και από νομικής απόψεως και από για λόγους πρακτικούς οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις συλλογικές συζητήσεις που γίνονται για τις διατάξεις που τους πλήττουν, που τους αφορούν σε τελευταία ανόληση ούτε σε κλαδικό επίπεδο, ούτε σε τομεακό επίπεδο, ούτε σε εθνικό επίπεδο κτλ. Άρα δεν εκπροσωπούνται οι άνθρωποι αυτοί σε οποιασδήποτε συλλογικές διαπραγματεύσει και συζητήσει. Και κάτι τι άλλο είναι προφανές πως ε, στα διάφορα κράτη-μέλη έγιναν τα τελευταία χρόνια προσπάθειες για να, να, προσ, να, να, να, προσαρμοστεί λιγάκι και το εργατικό δίκαιο και οι εργασιακές, εφόσον αλλάζουν σχέσεις. Αλλά ε, αυτά δεν έγιναν με τον σωστό, με τον ίδιο τρόπο παντού. Υπάρχουν πολλά κενά και ε, τα πράγματα δεν ε, απέδωσαν καρπούς. Τι λέμε τώρα, τι προτείνουμε. Να αναθεωρήσουμε κάποια νομικά πλαίσια αναφοράς. Παράδειγμα, υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις μαζικές απολύσεις σε περίπτωση αναδιάρθρωσης της επιχείρησης κτλ. Αλλά αυτή η νομοθεσία αφορά στους, σε αυτούς που είναι πλήρους απασχόλησης ή αορίστου χρόνου ή έκτακτη εργαζόμενοι ή οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου δεν καλύπτονται από αυτή την νομοθεσία. Ποια είναι η μοίρα λοιπόν αυτών των ανθρώπων, αυτών των μορφών εργασίας μετά από αυτό. Δεύτερο, δεύτερη πρόταση. Νομίζω ότι πρέπει να αναδιοργανωθούν κάποια επίπεδα κοινωνικού διαλόγου είτε σε επίπεδο επιχείρηση είτε σε επίπεδο τομέα είτε σε επίπεδο περιφέρειας δεν ξέρω ούτω ώστε να αλλάξουν λοιπόν οι οργανωτικές δομές ούτω ώστε να επιτραπούν να επιτραπεί η συμμετοχή στις συζητήσεις αυτών των εργαζόμενων και τρίτη πρόταση που κάνουμε, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι την σήμερα ημέρα ε, ε, συμβαίνουν σημαντικά πράγματα, σημαντικές αλλαγές με τους αυτοαπασχολούμενους και με τις τριγωνικές σχέσεις εργασίας. Μέχρι τώρα είχαμε διμερείς σχέσεις εργασίας, έτσι, το αφεντικό και ο εργαζόμενος. Ο, ο σήμερα η ημέρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι αποδημερείς και έχουν γίνει τριμερείς οι σχέσεις. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας να προσέξουμε αυτές τις μορφές εργασίες που αναδύονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και να προλάβουμε κάποια πράγματα. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω από τα πλούσια αυτά συμπεράσματα ότι η προηγούμενη Επιτροπή έκανε σκόπιμο να παρουσιάζεται και πάλι τις εργασίες στη νέα Επιτροπή, τόσο ώστε ο νομοθέτης που πρέπει να λάβει υπόψη ε, την πραγματικότητα των εξελίξεων στην αγορά εργασίας να είναι δεόντως ενημερωμένος. Λοιπόν, για να δούμε, να ακούσουμε τους ομιλητές μας, Αλεξάνδρες Σέρκας, η κυρία Σρέτερ, αρχίζουμε και βλέπουμε. Ο κύριος ε, Σέρκας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, την ε, παρουσίαση που έκαναν ε, οι δύο εισηγητές. Ελπίζω να έχω και χρόνο για να μπορέσω να μελετήσω και πολύ πιο διεξοδικά αυτή την αυτή τη μελέτη. Αν την έχετε στα ισπανικά ή στα γαλλικά θα την προτιμούσα από τα αγγλικά. Αλλά είναι σαφές ότι έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό έγγραφο στα χέρια μας. Και ε, εξίσου σημαντικό θα ήταν, επειδή δεν το άκουσα, να φανεί από αυτό το κείμενο ε, σαφώς ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός προβλήματος και δεν έχουμε λύση. Και χρειαζόμαστε νέες οδούς και νέα νομοθετικά μέσα προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα οικονομική πραγματικότητα, αυτή τη νέα ε, πραγματικότητα των εργασιακών σχέσεων που δεν έχει ε, και μεγάλη σχέση με τον τρόπο ε, που αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα τις συλλογικέ συμβάσεις εργασίας. Στην καρδιά λοιπόν του κοινωνικού εργασιακού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτές τις πτυχές. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον εξετάσατε επίσης και τις νομικές βάσεις που έχουμε στη διάθεσή μας εδώ στο Κοινοβούλιο για να εξετάσουμε το θέμα αυτό. Ε, έχουμε τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας, τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τα λάβατε αυτά υπόψη, είδατε τι νομικές δυνατότητες έχει το Κοινοβούλιο για να αντιμετωπίσει θέματα τα οποία προφανώς θα χρειαστεί να τα αντιμετωπίσει ε, πολύ σύντομα, διότι αν δεν τα έχετε μελετήσει αυτά θα βρεθούμε ενώπιον μια σκοτεινή κατάσταση ε, εργασιακού δικαίου στην Ευρώπη. Θα έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, δύο κατηγορίες εργαζομένων, αυτών που έχουν δικαιώματα και αυτών που δεν έχουν. Η κυρία Σρέντερ. Και μετά η κυρία Μωρό. Ε, ευχαριστώ πολύ. Όπως και ο συνάδελφος Σέρκας, <clears throat> θα ήθελα κι εγώ να θέσω ορισμένα ζητήματα. Πρώτο ερώτημα. Ε, επειδή μόλις τώρα πήραμε τη μελέτη, ποιοι ήταν οι τύποι εργασίες, ποιες ήταν οι μορφές εργασίας που μελετήσατε. είδατε μορφές εργασίας μόνο όπου ο εργαζόμενος εξαρτάται από κάποιον άλλον, είναι υπάλληλο αν θέλετε ή όχι. Το λέω αυτό γιατί είδαμε τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν εργαζόμενοι, κυρίως εργαζόμενες που είναι μεταξύ των, της φάσης του υπαλλήλου, αν θέλετε και του αυτοαπασχολούμενου. Είναι κάποιε ενδιάμεσε φάσεις. Πρώτο ερώτημα αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Τα συστήματα κοινωνική ε, προστασίας, κοινωνική ασφάλισης για τους εργαζόμενους. Πράγματι, δεν ξέρουμε πώς εφαρμόζονται για τις νέες αυτές άτυπες μορφές εργασίας. Ε, είπατε ότι είναι πρόβλημα αυτό. Απ' την άλλη μεριά ε, έχετε προτάσεις, δηλαδή ψάξετε να δείτε αν κάποιος κάνει ως αυτοαπασχολούμενος δύο-τρία επαγγέλματα. Ε, ένα-δυο στη χώρα και άλλο ένα στην άλλη μεριά των συνόρων, παραδείγματος κάνει μια άλλη, μια τρίτη δουλειά. Συνολικά τα κοινωνικά του επιδόματα είναι τα ίδια όπως αν δούλευε ε, πολύ μονίμως στην ίδια χώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μελέτη και ε, θα σχολιάσω τρία σημεία. Πρώτον, θα συμφωνήσω με τον κύριο Σέρκας που μας λέει ότι πρέπει να την αντιπαραβάλουμε στα ε, κείμενα που υπάρχουν ή να δούμε πού υπάρχουν κενά. Ε, στην προηγούμενη θητεία, στην Επιτροπή μας, ασχοληθήκαμε με την οδηγία για την προσωρινή εργασία και βλέπουμε εδώ ότι μπορούμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία πλήρωση των κενών, αλλά πρώτα πρέπει να τα εντοπίσουμε. Και μια τέτοια μελέτη, όπως αυτή μας παρουσιάστηκε, ακριβώς αυτό το στόχο έχει, να εντοπίσουμε τα κενά. Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ε, ε, οι ομάδες ε, έργου εργοδοτών ποια θέση έχουν. Τρίτον, υπάρχουν τομείς όπου αντίθετα μπορούμε να επιταχύνουμε εμείς τη διαδικασία. Ναι. Εννοώ ιδιαίτερα ότι έχει σχέση με την ε, φόρο ζωής κατάρτιση την... Ε, και βασιζόμενοι στις νέες τεχνολογίες ή στα φόρα κοινωνικού διαλόγου, μπορούμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία, να προσδώσουμε μια νέα διάσταση πολύ πιο σημαντική και πολύ πιο αποτελεσματική κατά τη γνώμη μου. στις παραδοσιακές ε, μορφές εργασίας. Μη βλέπουμε μόνο τα αρνητικά σημεία. Υπάρχουν και να, ναι. Υπάρχουν νέες μορφές που δεν αναφέρονται, για τις οποίες έχουμε ερωτηματικά και έχουμε και δυναμικό ε, επίσπευση στις διαδικασίες χάρη στις νέες τεχνολογίες για να ε, αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των νέων μορφών εργασίας. Σας ευχαριστούμε, κύριο Τόμας Μάν. <clears throat> Ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω κάτι για τη φλεξική flexicurity ουσιαστικά είναι θα έλεγε κανείς είναι κάτι καλό. Ο, έχουμε και τα δύο καλά. Απ' τη μια υπάρχει ευελιξία και τα λοιπά, απ' την άλλη μεριά υπάρχει και μια κάποια ασφάλεια. Ξέρω ότι η έννοια αυτή έχει ε, γίνει αντικείμενο επίθεση από πολλούς. Εγώ μάλιστα πίστευα και όλα ότι η, εγώ όμω πίστευα ότι η έννοια αυτή είναι αρκετά δυνατή. Ότι... Ε, μας δίνουν τη, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και το ε, την πίτα ολάκερη και το σκυλοχορτά, το φάλγα, εγώ δεν ξέρω. Ή, ε, ξέρω ότι κάποιες συνδικαλιστικές, οργα, συνδικαλιστικές οργανώσεις ε, είναι αντίθετες και αναρωτιέμαι γιατί τελικά έχουν ε, δεν έχουν περάσει και στους εργαζόμενους κάποιες θετικές ε, πτυχές της Flex Security. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και, δυν και ε, αδυναμίες αλλά και δυνατές τις πτυχές της έννοιας αυτής. Νομίζω, εσείς τι νομίζετε, γιατί πραγματικά νομίζω ότι δεν έχουμε ε, κατανοήσει όλοι σωστά την έννοια αυτή. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν το λόγο. Ο κύριο Χέντελ. Ευχαριστώ τώρα, το είπατε σωστά το όνομά μου. Μετά τον ε, κύριο Τόμας Μάν θα ήθελα να πάρω και εγώ το λόγο και να πω ότι ε, ένα από τα θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσει μια νέα μορφή εργασίας που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η λεγόμενη αυτό που λέμε στη Γερμανία Leiharbeit ε, δηλαδή ενοικίαση εργαζομένου έτσι ε, δανεική εργασία δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι η τι σημαίνει η έννοια αυτή. Πάντως οι άνθρωποι αυτοί πλήττονται σημαντικά από την κρίση και κατά πάσα πιθανότητα διατρέχουν τον κίνδυνο να ε, μην μπορούν να βρουν ε, εργασία στο μέλλον. Λέω λοιπόν ε, ότι αυτή το Προεδρείο της Επιτροπής μας θα πρέπει να ασχοληθεί λιγάκι και με το θέμα αυτό να αντιμετωπιστούν τα κενά που υπάρχουν, να συμπληρωθούν στο βαθμό που μπορούν τα κενά αυτά και να προσπαθήσουμε να εισάγουμε κάποιους κανόνες σχετικά με αυτήν τον τύπο εργασίας. Ωραία λέει η Πρόεδρος. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο μελετητές θα πάρει πρώτο το λόγο. Σίγουρα τη μελέτη αυτή δεν ξανασυζητήσουμε, η κομμάτια της μελέτης αυτής που δεν είναι λόγο θεωρώ ότι σήμερα είναι η τελευταία φορά που κουβεντιάζουμε το, τα θέματα αυτά. Θα έχουμε και καινούριο επίτροπο την επόμενη φορά, οπότε σίγουρα τα ξαναπούμε. Θα αρχίσω εγώ απαντώντας και θα συμπληρώσω ο συνάδελφος. Θα είμαι σύντομος, πάρα πολύ σύντομος. Λοιπόν, απαντώ. Ναι, ε, πολλά κράτη-μέλη συζητούν το θέμα ε, αφενός των ε, αυτοαπασχολούμενων αφετέρου των μισθωτών με επιλογές προς το παρόν που ακολουθούν διαφορετικές κατευθύνσεις. Φερρυπίν, κάποια κράτη-μέλη έχουν εισαγαγή, τώρα εισάγουν μια τρίτη κατηγορία Ισπανία, παραδείγματο χάρη, με το καθεστώ των αυτόνομων εργαζομένων, το Λουξεμβούργο, έχουν εντελώ ε, αρνηθεί να ασχοληθούν με το ζήτημα. Αλλά είναι πήγον το πρόβλημα σε όλα τα κράτη-μέλη τη σήμερον ημέρα και δεν υπάρχει προς το παρόν ενιαίος ευρωπαϊκός ορισμός της λέξης εργαζόμενος. Το δεύτερο θέμα που σχολιάσατε είναι αυτές οι ομάδες, οι ενώσεις των εργοδοτών. Δεν προκύπτει αυτό άμεσα από την έκθεσή μας, γιατί ε, ε, παρατηρείται αυτό σε κάποια κράτη-μέλη, Γαλλία, Βέλγιο και κάποια άλλα. Δεν έχει τέτοια ευρωπαϊκή εμβέλεια ώστε να ε, κρίνουμε σκόπιμο να το συμπεριλάβουμε στα συμπεράσματά μας. Παρ' όλα αυτά δεν ε, παραγνωρίζουμε το ότι σημειώνεται το φαινόμενο σε κάποια κράτη-μέλη. Πιο ικανοποιητική απάντηση δυστυχώ δεν έχω. Τρίτο θέμα και μετά θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου. Είναι η νομική ε, ικανότητα. Μπορώ να απαντήσω από διάφορες, ε, από διάφορα εφαλτήρια αν θέλετε. Ε, έχει προκύψει και σε προηγούμενες συζητήσεις αυτό το θέμα. Ναι, το θέμα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία μας προσφέρει μια νομική βάση ούτω ώστε να επιτύχουμε ε, σε ένα ορισμένο βαθμό μια ισότιμη μεταχείριση και την ε, συναφή προστασία. Αυτό είναι ένα εφαλτήριο στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε και να δώσουμε απάντηση. Δεύτερη προσέγγιση, αν θέλετε, είναι ότι η αναθεώρηση, η αναθεώρηση και το τονίζω αυτό της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να επιτρέψει όπως ε, για την ε, νομοθεσία για τις ε, μαζικές απολύσεις, μπορεί να μας επιτρέψει να αναθεωρήσουμε την νομοθεσία για να λάβουμε υπόψη τις νέες μορφές εργασίας. Θα είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί για τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης, φυσικά. Για τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης το γνωρίζετε, είναι πολύ πιο αδύναμη η νομική βάση. Ένα, δύο, ε, σημειώσαμε το πρόβλημα, προς το παρόν δεν έχουμε πολλές λύσεις να προτείνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δίνω το λόγο στον συνάδελφο να απαντήσει στα υπόλοιπα ερωτήματα. Πολύ σύντομα. Στα θέματα των προβλημάτων της κοινωνικής ασφάλισης, ε, φυσικά και έχετε δίκιο τα προβλήματα της κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως όσον αφορά στην εναρμόνιση των διαφόρων νέων μορφών εργασίας, των νέων μορφών συμβάσεων, είναι ε, κάτι το οποίο σαφώς πρέπει να επιλύσουμε, διότι είναι και τεχνικώς πολύ δύσκολο. Να σας ε, πω για παράδειγμα το θέμα το διασυνοριακό και μόνο πόσες δυσκολίες θα δημιουργήσει. Ε, έχουμε διαφορετικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία είναι πολύ περίπλοκο ε, και υπάρχουν και προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την οδηγία ε, για τη διαμεθοριακή εργασία. Τώρα, η ευελικτή ασφάλεια. Σαφώς είναι ένα συνδυασμό στοιχείων, σωστά το ορίσατε εσείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό και κατανοητό το πώς είναι το θέμα γενικώ, αλλά το θέμα είναι η εφαρμογή από εκεί και πέρα. Κανείς ε, σχεδόν στα κράτη-μέλη δεν λέει σήμερα ότι η ασφάλεια... είναι κάτι το οποίο έχει εγκριθεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται σταδιακά και μέσω της διαδικασίας της Λισαβόνας και των οδηγιών απασχόλησης, αλλά δεν υπάρχει και ένα πανευρωπαϊκό φόρουμ ε, συζήτησης για να έχουμε ε, ευελιξία και ασφάλεια στην εργασία συντονισμένα, γιατί εξακολουθεί να είναι ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών η εφαρμογή της νομοθεσίας. Εγώ σας έδωσα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά ε, συνήθως όταν θέλουμε να μεταφέρουμε τις κοινέ αρχές της ε, ευελικτασφάλειας, ε, Είδαμε ότι υπήρχαν κάποια κράτη-μέλη που έκαναν πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις λαμβάνοντας υπόψη μόνο την ευελιξία και ξεχνώντας την ασφάλεια. Θα πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να γίνεται μια ισορροπημένη εφαρμογή και μάλιστα θα πρέπει να παρακολουθείτε, να αποπτεύετε από ε, όργανα τα οποία θα είναι ανεξάρτητα και θα μπορούν να παρακολουθήσουν και να έχουν όχι μόνο μια ισορροπία αλλά να έχουν και μια προσαρμογή ε, στις ανάγκες του σήμερα. Υπάρχουν για παράδειγμα μέτρα τα οποία εγκρίνονται τώρα λόγω της κρίσης ε, στα οποία δεν υπάρχει πάντα κατάλληλη ισορροπία. Οι κοινωνικοί εταίροι ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάστηκαν αρκετά, έχουν διαμορφώσει την άποψή τους και έχουν λάβει υπόψη τους το θέμα της ευελικτασφάλειας, ε, θέλησαν να υπάρχει ευέλικτη εφαρμογή. Η ευελιξία ούτως ή άλλως έχει να κάνει και με τις δυναμικές που διαπιστώνουμε. Οι δυναμικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σήμερα έχουν να κάνουν με την αύξηση της παραγωγικότητας, της αύξησης της παραγωγικότητας των επιχειρώσεων. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το πώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένα, ε, ότι θα έχουμε ένα κοινωνικό σύστημα ευρωπαϊκό το οποίο θα προσαρμόζεται στους καιρούς μας. Και τέλος, η ερώτηση του συντονιστή για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτή τη στιγμή δεν ε, ασχοληθήκαμε με τις βάσεις που θα μπορούσε να περιλαμβάνει η, στρατηγική της, η συνθήκη της Λισαβόνας συγγνώμη, για, την, ε, ε για την εφαρμογή για τις άτυπες μορφές εργασίας, αλλά Έχουμε λάβει υπόψη την έννοια των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα βασικά εργασιακά δικαιώματα έχουν αρκετά νομικά κολλήματα και φυσικά αυτό λήφθηκαν υπόψη. Ε, λάβαμε υπόψη μας ε, κυρίως διεθνείς και πολυμερείς πτυχές, αλλά υπάρχουν για παράδειγμα τα core labor rights, τα βασικά εργασιακά δικαιώματα που αποτέλεσαν το βασικό, το ελάχιστο, ένα κατόφλι από το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε ε, κάποιες βασικές εργασιακές αρχές στην Ευρώπη. Εμείς ε, αναλύουμε εις βάθος ε, τι μπορούμε να έχουμε από εκεί και πέρα και έχουμε πέντε βασικά στοιχεία τα οποία θεωρούμε ότι θα ήταν μια καλή προσέγγιση από πλευράς κοινοτικού και εκτιμένου ε, για τα βασικά εργασιακά δικαιώματα. Καταρχάς τα ίδια τα συμβατικά δικαιώματα. Δεύτερον, τα δικαιώματα που σχετίζονται με την απασχόληση και την αγορά εργασίας. Για παράδειγμα υπάρχουν ε, δικαιώματα τα οποία σχετίζονται με την ευελικτασφάλεια και έχουν να κάνουν και με μετάβαση από δουλειά σε δουλειά, job to job transitions ή για παράδειγμα τη μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας ή από, αγορα... από εργασία σε εργασία. Ένα τέταρτο στοιχείο είναι τα ε, ε, στοιχεία τα οποία επιτρέπουν να ασκεί κάποιος αποτελεσματικά τα δικαιώματά του και το πέμπτο στοιχείο είναι τα συλλογικά δικαιώματα, τα δικαιώματα εκπροσώπησης και συμμετοχής. Με αυτές τις πέντε κατηγορίες, οι οποίες φυσικά η κάθε μία έχει διαφορετική εθνική προσέγγιση, θα μπορούσαμε να οικοδομήσουμε και να μελετήσουμε ποια θα είναι η νομική βάση στις συνθήκες, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια κάποια ισορροπία. Ευχαριστώ πολύ για μια πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής είναι πάρα πολύ καλή στιγμή στην οποία έγινε η παρουσίαση αυτής της έκθεσης. Νομίζω ότι μπορούμε να